Συναγαπητοί uh, συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίστε, διότι πρόκειται να αρχίσουμε. Hm? Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας με μικρή καθυστέρηση. Ο Επίτροπος ξέχασε τα γυαλιά του και εφόσον δανείστηκε τα γυαλιά κάποιου άλλου, δεν ε, και ένα άλλο αστείο, δεν πρόκειται να σας το μεταφέρω. Οποιοδήποτε λάθος κάνει ε, δεν θα έχει να κάνει με την παρουσίασή του. Είναι ανθρώπινος ο Επίτροπος. Οπότε και εγώ δεν θα φορέσω τα γυαλιά μου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Επίτροπος, Βεβαίω, εμεί έχουμε πέντε επιτρόπους, όπω ανακαλύψαμε κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, αλλά είναι ο ε, αποκλειστικό αρμόδιο για την εσωτερικέ υποθέσει είπε ότι θα έρθει να μας επισκεφτεί το συντομότερο δυνατόν και κράτησε την υπόσχεσή του. Ήταν συνεχώς σε επαφή, μπορώ να το διαβεβαιώσω, από την ακρόαση. Θα ήθελα αυτό να σημειωθεί, ότι εξετάζει συνεχώς το χαρτοφυλλοκιά μας από την ημερομηνία της ακρόασης και έρχεται σήμερα εδώ ήταν σε συνεχή επαφή μαζί μας και με το προσωπικό μας και είμαι ευγνώμων γι' αυτό χτες. Όπως θα σας το πει, είχαμε μια συνάντηση μεταξύ των Πρόεδρων όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και επιτρόπων και μπορώ να σας πω ότι τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων είναι το δικό μας χαρτοφυλάκιο, θεωρήθηκε από τα βασικά χαρτοφυλάκια του Σώματος των Επιτρόπων, ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς, κατέστησε σαφές ότι η μετανάστευση και άλλα τέτοια θέματα θα έχουν ε, μεγάλη προτεραιότητα. Γι' αυτό χαιρετίζουμε εδώ την παρουσία του Δημήτρη Ευραμόπουλου. Εξ ονόματος της Επιτροπής θα μας μιλήσει 10-15 λεπτά και μετά θα έχουμε τον πρώτο γύρο από τους συντονιστές και μετά όλα τα μέλη θα μπορούν να λάβουν απαντήσεις δεν θα είναι η μόνη συνάντηση με τον Επίτροπο, είναι μέρος της διαδικασίας, ε, θα μιλήσει για τα πάντα, θέλουμε και εμείς ε, να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά θα ήθελα να μιλήσει για τα βασικά του θέματα, τα βασικά, τα πιο σημαντικά θέματα, να μην υποκύψει στον πειρασμό να μιλήσει για όλα ας μιλήσει για τα θέματα αυτά, τα πιο βασικά, τα πιο σημαντικά, διότι θα έρχεται τακτικά να μας επισκέπτεται. Κύριε Επίτροπε, σας δίνω τον λόγο. Σας παρακαλώ να κάνετε την πρώτη σας δήλωση στην Επιτροπή και μετά θα δεχτείτε ερωτήσεις από τα μέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αλλά φόσον κάνατε ε, σχόλιο περί ανθρωπιάς σε αυτήν την Επιτροπή δεν μπορεί κανείς παρά να είναι ανθρώπινος. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτον να σας πω ότι αισθάνομαι τιμή και μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Οι πρώτες τέσσερις εβδομάδες από το ανέλαβα αυτή τη θέση ήταν πάρα πολύ φορτωμένες. Το ομολόγο την περασμένη εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, είχα το, το μπάπτισμά μου της Ολομέλειας ε, πήγα σε σημαντικές συναντήσεις για να δώσω τις κατευθυντήριες πολιτικές γραμμές για βασικά θέματα και για το πρόγραμμα WELF για το επόμενο χρόνο για να δούμε την στρατηγική ε, για τους βασικούς φακέλους που έχουμε. Θα αναφερθώ σε ένα μέρος της εργασίας που έγινε στην ομιλία μου. Θα ήθελα να αρχίσω με το θέμα της μετανάστευσης μαζί με την το Προεδρείο Είχαμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψει στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Θα ήθελα να εκφράσω την ευχαριστίες μου σε όλους σας ε, για καρποφόρο συζήτηση και επικοδομητική κυρίως ε, σχετικά με το, την σημασία των μεταστευτικών πιέσεων ε, της οδούς, ασφαλής οδούς για τους ετούντες άσυλο και την συνεργασία με τρίτες χώρες σημείωσα προσεκτικά τις παρεμβάσεις σας. Σχετικά ε, με την κατάσταση που υπάρχει σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ε, που συμφωνήθηκαν από την Task Force ε, Μεσογείου και του Συμβουλίου του Οκτωβρίου, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω σε ένα scorecard το οποίο μοιραστήκαμε μαζί σε μια κάρτα βαθμών και μετά θα απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Έχω ε, την πρόθεση να συνεχίσω στο δρόμο αυτό και περιμένω το ψήφισμά σας μετά τη συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τη δράση μας για να αντιμετωπίσουμε τους ε, λαθρεοδιακινητές που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών. Αυτή από τις προτεραιότητες μου για να προλάβουμε περαιτέρω απώλεια ζών. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή αναπτύσσει ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε ε, την, ε, την λαθρέα διακίνηση και να διαφυλάξουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των μεταναστών ανεξάρτητα από τη θέση τους. Είναι τα μέτρα που διευκρίνησα στην παρέμβασή μου στην διαδικασία της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που είχε ως θέμα την μετανάστευση και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Λαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλίες για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την δίωξη των εγκληματιών με κοινέ δράσεις με την υποστήριξη της Europol. Αλλά εάν θέλουμε πραγματικά βιώσιμες λύσεις, οι προσπάθειες αυτές πρέπει να είναι μέρος ολοκληρωμένης προσέγγισης, όπου η δράση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνοδεύεται με ενισχυμένη συνεργασία με τρίτες χώρες. Ένα σαφές παράδειγμα ολοκληρωμένης προσέγγισης είναι η διαδικασία Καρτούν που άρχισε την περασμένη εβδομάδα στη Ρώμη. Η διαδικασία είναι καλό παράδειγμα για το πώς κανείς να έχει ένα διάλογο με τρίτες χώρες βάσει κοινή εμπιστοσύνη. Ε, με ε, συγκεκριμένα προγράμματα και χρηματοδοτικούς πόρους. Ε, ήταν πρώτη φορά που θέσαμε επιτάπητο στο θέμα αυτό οι χώρες προέλευσης, οι χώρες διάλευσης και οι χώρες προορισμού. Στα πλαίσια της διαδικασίας θα χρηματοδοτήσουμε τα πρώτα πρόγραμμα προς όφελος των μεταναστών ε, που έρχονται από την Ανατολική Αφρική επιπλέον. Ε, πόροι έχουν διοχετευθεί για την βοήθεια και ενίσχυση της συνεργασίας με τους Αφρικανούς εταίρους για την καταπολέμηση της, του λαθρεμπορίου, της λαθρέας διακίνησης. Ήθελα να σας πω ότι στη Ρώμη οι συναντήσεις ήταν πολιτικά πολύ σημαντικές, όχι μόνο επειδή κατορθώσουμε να φέρουμε στο ίδιο διαπραγματευτικό τραπέζι χώρες όπως την Ερυθρέα και την Αιθιοπία, αλλά επειδή είχαμε και τη δυνατότητα να ακούσουμε τις απόψεις των Αφρικανών ομολόγων μας. Όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση, επαναλαμβάνω τη δέσμευσή μου να έχουμε μια νέα πολιτική για την νόμιμη μετανάστευση να γίνει βασική μου προτεραιότητα. Μια επιτυχημένη τέτοια πολιτική θα είναι βασική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και προστασία του κοινωνικού μας μοντέλου. Όπως τόνισα, στην διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι για την νόμιμη μετανάστευση πριν από δύο μέρες, η ε, νομιμοποίηση, οι καμπάνιες εκστρατείες νομιμοποίησης είναι μια αντίδραση μεταξύ άλλων θα πρέπει να υπάρχουν ε, για να μην υπάρχει αβεβαιότητα μεταξύ των μεταναστών ε, που θεωρούν ότι η νομιμοποίηση είναι κάτι το απρόβλεπτο. Θα πρέπει να εστιαστούμε στο να δημιουργήσουμε άλλες νόμιμες οδούς. Για να εκπονήσουμε αυτήν την πολιτική θα εργαστούμε στενά με τις επιχειρήσεις, με τις μικρές επιχειρήσεις, τα συνδικάτα και ε, τα ενδιαφερόμενα ε, μέλη αυτού του Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα. Η δέσμευση των οικονομικών ενδιαφερομένων είναι πάρα πολύ σημαντική για να αλλάξουμε τη ρητορία περί μετανάστευσης που είναι προϋπόθεση για την επιτυχία και τον αντίκτυπο των αλλαγών πολιτικής στον τομέα αυτών. Βασίζουμε επίσης στην πολύτιμη πολιτική σας υποστήριξη θα αρχίσουμε εξετάζοντας τις υφιστάμενες πολιτικές όπως την μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσα να γίνουν πιο ελκυστικές και αποτελεσματικές αυτές οι πολιτικές. Ένα νέο στοιχείο της νέας πολιτικής είναι η ε, ε, αναδιατύπωση των οδηγιών περιερευνητών και φοιτητών. Έχουμε κάνει φιλόδοξη πρόταση για κανόνες πιο ελκυστικούς, πιο ενδιαφέροντες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ισχυρή υποστήριξη στην πρότασή μας. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα εκφράσει μια κοινή θέση, αλλά η Ιταλική Προεδρία κατόρθωσε να προωθήσει τη συζήτηση σε σημαντικό τομέα όπως την κινητικότητα και μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι στο τέλος του έτους το Συμβούλιο θα έχει ε, συμφωνήσει την εντολή αυτή. Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας της πρότασής μας και εδώ βασίζουμε και πάλι στην ε, συνεχή σας υποστήριξη για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι οι περισσότεροι μετανάστες που έρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Ένωσης έρχονται για λόγους εκτός της απασχόλησης. Επανένωση, η οικογενειακή είναι σημαντικότερη κατηγορία με μεγάλο αριθμό ε, που λαμβάνουν ε, θεωρήσεις παγκόσμιας προστασίας και για ανθρωπιστικούς λόγους. Τα άτομα αυτά έρχονται με τη μόρφωσή τους και τις προσόντα τους είναι προς όφελος των χωρών μας να συμβάλλουμε ούτως ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ικανότητες τους. Η ένταξη στην αγορά εργασίας των νομίμων μεταναστών είναι ένας τομέας όπου όλο και περισσότερο θα εργαζόμαστε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναζητήσει την γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την Συμφωνία PNR μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, τα στοιχεία των επιβατών. Περιμένουμε την γνωμοδότηση, την απόφαση του δικαστηρίου. Η Επιτροπή πιστεύει ότι θα δώσει τη σαφήνεια που απαιτείται το δικαστήριο για να προχωρήσουμε με τη συμφωνία αυτό, διότι σε όλους τους επιβάτες ε, δίδονται, έτσι παρέχονται πρόσθετα δικαιώματα. Κατά την άποψη της Κομισιόν, η απόφαση την περασμένη εβδομάδα δεν έχει αντίκτυπο πάνω στην ουσία ή πάνω στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για την οδηγία PNR στοιχείων επιβατών. Υπάρχουν τρία σημεία ακόμα ε, τα οποία ε, εκκρεμούν ε, η αναγκαιότητα του σχεδίου PNR, το πακέτο προστασίας δεδομένων που είναι υποδιαπραγμάτευση και η απόφαση περί διατήρησης στοιχείων PNR που είναι κάτι το διαφορετικό. Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την, τα επιχειρήματα της πρότασης. Χρειάζεται μια τέτοια συμφωνία για να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων των ατόμων που ζουν στην Ευρώπη. Μερικοί από εσά έχουν ακόμη αμφιβολίες για την αναγκαιότητα της διαδικασίας αυτής του PNR. Όπως είπα στον πρόεδρο, είμαι έτοιμος να διευκολύνω τους εμπειρογνώμονες που θα μας δώσουν ε, με πραγματικά ε, παραδείγματα πώς ε, τη διαδικασία PNR είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας και για να απαντηθούν οι ερωτήσεις των μελών. Θα είναι χρήσιμο να έχουμε μια τέτοια παρουσίαση όσο το δυνατόν συντομότερα λόγω της αναγκαιότητας για την ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα φορτόχρονα της ανάγκης να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση του θέματος, η Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα και να ε, προκαταλάβουμε τα διάφορα ε, στοιχεία που θα μπορούσε το πακέτο να εισαγάγει όταν τεθεί σε ισχύ. Η Επιτροπή πιστεύει ότι υπάρχουν ορισμένες αλλαγές που θα πρέπει να εισαχθούν στην πρόταση PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει μια μεγαλύτερη προστασία ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων και για να βεβαιωθούμε ότι η πρόταση συνάδει πλήρως με την απόφαση περί διατηρήσης στοιχείων. Να ενισχύσουμε την εποπτεία ε, πάνω στις ε, μονάδες πληροφοριών που είναι υπεύθυνε για την διαδικασία δημιουργώντας ε, έναν ε, ρόλο, μία θέση για έναν ανεξάρτητο αξιωματούχο. Επίσης, με την μονάδα, η συνεργασία με την μονάδα συνεπάγεται ότι τα άτομα θα είναι εκπαιδευμένα, το να ε, πρέπει να έχουμε περισσότερο μέτρα προστασίας και να δώσουμε στην Κομισιόν δύο χρόνια αντί για τέσσερα να αναθεωρεί την οδηγία λειτουργίας και να αναφέρει στο Κοινοβούλιο. Είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε με το ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να υπάρξει πρόοδος στο θέμα του PNR. Βεβαίως θα προτείνετε τροπολογίες ε, για να βελτιωθεί η πρόταση αυτή. Και καλό σας καλό και σας ενθερίνω να το πράξετε. Και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας ε, πάνω στο θέμα αυτό. Η θα υποστηρίξει τις προσπάθειες ούτως ώστε η πρόταση να είναι πιο ισχυρή από την άποψη των εγγυήσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε την εργασία για το PNR. Πολλά κράτη-μέλη έχουν τα δικά τους εθνικά συστήματα, το γνωρίζετε αυτό. Εμείς ε, παρακολουθούμε εκ του σύνεγγες τις προσπάθειες αυτές, ούτως ώστε η εργασία αυτή να μην επηρεάζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών μας, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Δεν θέλω να επανέλθω στο ίδιο θέμα σχετικά με την χρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων PNR. Η Κομισιόν έδωσε σαφή απάντηση και θα ήθελα να το σημειώσετε αυτό ακόμη και χωρίς χρηματοδότηση μερικά κράτη-μέλη προχωρούν μερικά του συστήματα PNR. Ελήψη ευρωπαϊκών κανόνων για το PNR κινδυνεύουμε να έχουμε αποκλίνοντα συστήματα τελείως διαφορετικά, με διαφορετικά επίπεδα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε ένα πανευρωπαϊκό σχήμα. Επιπλέον, η Κομισιόν θα οργανώσει τον Ιανουάριο μια συνάντηση μεταξύ των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων PNR και εκπροσώπων των Εθνικών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των αρχών αυτών. Εν κατακλείδη, θα πρέπει να λάβω υπόψη την βούληση όλων των συνομοθετών. Γι' αυτό απευθύνομαι σε εσά, κάνω έκκληση σε εσά. Είναι θέμα ρεαλιστικής επιλογής μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί για να βελτιώσουμε ουσιαστικά την υφιστάμενη πρόταση και να εξασφαλίσουμε υψηλή προστασία για τους πολίτες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα μερικά λόγια για την διατήρηση των στοιχείων. Η παλιά οδηγία ε, διατήρησης δεν υπάρχει, αλλά ε, αυτή για τις τηλεπικοινωνίες είναι κρίσιμη για να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε σοβαρά εγκλήματα και τρομοκρατία. Χρειαζόμαστε λοιπόν να προβληματιστούμε για μια πολιτική που θα εγγυάται ταυτόχρονα την πλήρη τήρηση των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια των πολιτών και καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η νέα Επιτροπή θα εξετάσει και υπόσχεται τις καλύτερες επιλογές για το μέλλον ως προς την ε, διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα θέματα που συνεπάγεται αυτό. Εδώ η απόφαση ε, για την οδηγία είναι ο οδηγός μας ε, για να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για αυτό το οποίο γίνεται σχετικά με το πρόβλημα των ξένων μαχητών. Εργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να αναπτύξουμε μια κοινή προσέγγιση για την καλύτερη ε, χρήση ε, βάσει των ε, των εγγράφων που έχουμε για να έχουμε ελέγχου στα άτομα και ελέγχου στα έγγραφα. Η Κομισιόν προτίθεται να, να ε, δώσει κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, για το μέλλον και συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να έχουμε μέτρα αποτελεσματικά σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Schengen. Αυτά τα μέτρα θα επιτρέπουν ταχύτερη και βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών για ορισμένες επισημάνσεις σχετικά με ξένους μαχητές. Ε, τώρα ε, θα ήθελα ε, τώρα να μιλήσω για τα έξυπνα σύνορα. Το, το, η Κομισιό θα παρουσιάσει μια νέα πρόταση και παράλληλα θα αποσύρει το νομοθετικό πακέτο του 2013. Το δεύτερο, η φάση ελέγχου, του Proof of Concept θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο 2015. Η Κομισιό θα ήθελε να παρουσιάσει τις νέες προτάσεις μετά στο τέλος του 2015 ή αρχή του 2016. Αυτή η αναθεώρηση θα ανταποκριθεί στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να εξασφαλίσει τα έξυπνα σύνορα. Η συμβολή του Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη των έξυπνων σύνορων είναι κάτι το κλειδί για την παρούσα ανασκόπηση. Θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας και κυρίως με τους δύο εισηγητές, τη Μαντάμ, Γυρια Ταγιό και τον κύριο Τεντιέ Στεχέρα. Ελπίζω ότι θα συμμετάσχω στην ακρόαση που προγραμματίζεται με τα Εθνικά Κοινοβούλια στο τέλος του Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, επιστολή που μου απευθύνατε καλώντας με σε τριμερή συνάντηση ε, για τις 9 Δεκεμβρίου. Αλλά δεν υπερβάλλω όταν σας λέω ότι δυστυχώς το ε, πρόγραμμά μου είναι ε, γεμάτος. Στις 9 πρέπει να είμαι στη Γενέβη για σημαντική διάσκεψη ε, για την επανεγκατάσταση των σύρων προσφύγων και στις 10 ε, εμείς όλοι οι επίτροποι πηγαίνουμε στο Λουξεμβούργο μετά την συνάντηση για την ορκομοσία. Προτείνω βεβαίως να λάβει χώρα η συνάντηση, διότι είναι σημαντική και πρέπει να λάβει χώρα πριν από τη συνάντηση της Κορεπέρο. Ο Γενικός Διευθυντής μου θα με εκπροσωπήσει. Έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να σας δώσει κατευθυντήριες γραμμές ε, για την δεύτερη φάση του Proof of Concept. Η Κομισιό έχει το πλήρες δικαίωμα πρωτοβουλίας, αλλά πρόθεσή μας είναι να εργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και όπως αναφέρατε στην επιστολή σας, εξακολουθούμε βεβαίως να περιλαμβάνουμε τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ο πρώτος μήνας ήταν σκληρός πολλά πράγματα είχαν ήδη δρομολογηθεί πριν αναλάβω τη θέση αυτό. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα ήθελα να πολλαπλασιάσουμε τις επαφές με μέλη του Κοινοβουλίου για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και φακέλους και να είμαστε σε συνεχή επαφή με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είχα την, ήθελα να αρχίσω στο Στρασβούργο αλλά δυστυχώς είχα να ασχοληθώ με την ατζέντα της Ολομέλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχετε δημιουργήσει μεγάλη συμπάθεια με το γεγονός ότι ξεχάσατε τα γυαλιά σας. Έχουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει στο παρελθόν ένα, έχει ένα ρεκόρ σε σχέση με το παρελθόν. Όλοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Κάποιος μου έστειλε SMS ότι θέλει να μιλήσει και δεν έχει έρθει κιόλας εδώ. Ίσως τα μέλη του προσωπικού του θα μπορέσουν να μιλήσουν στη θέση του. 26. Μα δεν έχουμε 26. Μέλη καν εδώ παρόντα. Είναι μια παράξενη κατάσταση λοιπόν. Πιο πολλοί θέλουν να μιλήσουν από ότι είναι παρόντες. μετά από τέσσερα χρόνια ίσως μπορεί να έχει αδειάσει τελείωση η, η από μέλη της Επιτροπής μας. Εν πάση περιπτώσει μάλλον δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε στις 5 γιατί μακρηγόρησε λίγα και ο κύριος Επίτροπος, 20 λεπτά δεν μπορούσα να τον εμποδίσω φυσικά. Παρακαλώ στους συναδέλφους να παραμείνουν στα δύο λεπτά. Ξεκινώ με τους συντονιστές, τρία λεπτά ίσως οι συντονιστές. και ξεκινώ με το ΕΛΚ, αλλά παρακαλώ δείξτε αυτοσυγκράτηση, μην δοκιμάστε να εγείρετε όλα τα ζητήματα τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσει σε όλα αυτά ο κύριος Επίτροπος. Ξεκινώ με την κυρία με τη Ρομπέτα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπατε πραγματικά σεβαστεί κατά αυτά που είπατε και στην ακρόασή σας ότι θα παραμείνετε σε επαφή με την Επιτροπή μας. Για την μετανάστευση. Για τη μετανάστευση το, τα θέματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για μας. Διότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε απομονωμένο, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν ολιστικό τρόπο. Εάν δεν υπάρχουν ε, ολιστικές στρατηγικές που να αντιμετωπίζουν όλες τις πτυχές του προβλήματος της μετανάστευσης, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον σκοπό μας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην, ε, στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή είναι άμεσο αποτέλεσμα των όσων συμβαίνουν στην υποσαχάρια Αφρική. Όμως η απάντηση δεν θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε ένα οχυρό Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, να αντιμετωπίσουμε τα κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος που εκμεταλλεύονται τους ε, ε, ευάλωτους και ευαίσθητους ε, αυτούς ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν έτσι ώστε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την φρικτή κατάσταση. Αυτά είναι επομένως ευρωπαϊκά θέματα τα οποία απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις. Τώρα, ποιε είναι οι ενέργειε, ποιε είναι οι δράσει που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε. Ε, θίξατε κάποιε από αυτέ. Η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να ε, εντείνει, να ενδυναμώσει τις, την, την αντιμετώπιση αυτών των παράνομων διακινητών. Η Frontex και άλλε υπηρεσίε θα έχουν στη διάθεσή του κάθε δυνατό μέσο για να μπορέσουν να κάνουν ε, το έργο του. Για το PNR άκουσα με ικανοποίηση αυτό που είπατε ότι η απόφαση που, που ελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα ε, για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Καναδά δεν θα επηρεάσει επί της ουσίας τις διαπραγματεύσεις για την οδηγία PNR. Ε, και άλλοι συνάδελφοι θα θίξουν το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η οδηγία αυτή θα αυξήσει, αν θέλετε, την, τα επίπεδα ασφάλειας και ε, θα υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι, κάτι το οποίο θα είναι ε, υπέρ της ασφάλειας όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ε, Μάλτα έχουμε κάποια ανησυχητικά νέα όσον αφορά την συμφωνία ανάμεσα στις αρχές της Μάλτας και την Κομισιό για την χορήγηση υπηκότητας. Υπάρχουν άτομα τα οποία αγοράζουν διαβατήρια και δεν, δεν γίνεται σεβαστή η προϋπόθεση του ενός χρόνου παραμονής στην διαμονή στην, στην Μάλτα. Ελπίζω η Κομισιόν να το ερευνήσει αυτό. Ευχαριστώ, Ρομπέρτα. Η... σεβαστή τα τρία λεπτά και οι υπόλοιποι συντονιστέ να σεβαστούν τα τρία λεπτά, παρακαλώ, για του ε, σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αβραμόπουλε. Το θέμα της μετανάστευσης. Πράγματι έχει πολλές απόψεις, ένα πολυεδρικό θέμα. Ελπίζω ότι μαζί μας θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε την ελευθερία διακίνησης της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των επιθέσεων που εκπορεύονται από διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης όμως να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε και το δικαίωμα για ατομικό δικαίωμα ασύλου πρέπει οποιαδήποτε λύση υλοποιήσουμε να εξασφαλίσει ότι οι πρόσφυγες θα έχουν τη δυνατότητα με ασφαλή τρόπο να έρθουν να υποβάλουν το αίτημά τους για άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η μετανάστευση μέσα στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ βρίσκω ενοχλητικό να υπάρχει η, στην επικεφαλίδα με την, ε, μαζί με τη μετανάστευση και το εμπόριο ανθρώπων. Το εμπόριο ανθρώπων είναι μια δράση κλιματικών οργανώσεων. Εγώ θα ήθελα να το θέσω αυτό μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και όχι να το συνδέσω με την ε, μετανάστευση γιατί αυτό οδηγεί σε συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν ε, ευχάριστο χαρακτήρα μεταξύ του πληθυσμού. Επίσης το θέμα των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αναλαμβάνονται για την ασφάλεια, εγώ ενοχλούμαι για το γεγονός ότι τα εθνικά συστήματα PNR οδηγούν σε, διακρί... σε διακρίσεις σχέση με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το αξιοσημείωτο, γιατί όλα τα κράτη-μέλη έχουν προσυπογράψει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις βασικές μας αξίες. Με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει η προστασία αυτών των δικαιωμάτων επί τη βάση εθνικών κανόνων και να είναι τόσο διαφορετική από το ένα κράτο στο άλλο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, τη βδομάδα αυτή, είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει μια μεγαλύτερη διευκρίνηση για το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει μια πολυπληθώρα μέτρων σε σχέση με τα θέματα ασφαλείας, αλλά βλέπουμε πάντα σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και σε επίπεδο εθνικό όλα αυτά τα μέτρα που έχουν σαν στόχο να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα δεν έχουν μία ε, σύνδεση μεταξύ τους και δεν συναρμόζονται σωστά. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα μπορέσουμε να δράσουμε αντί να έχουμε νέα μέτρα, να έχουμε μια μεγαλύτερη συνεργασία στα θέματα αυτά. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν μπορούσατε να μου πείτε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια νέα ε, διευκρίνηση σε σχέση με μια νέα συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα πιενά, να μου πείτε τι γίνεται και με το πακέτο για την προστασία των δικαιωμένων, πώς θα εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση για την φύλαξη των προσωπικών δεδομένων. Εγώ ξέρω ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το θέμα των λεγόμενων foreign fighters όταν δεν έχουν πραγματική λειτουργία του συστήματος αυτού. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Κίρκοπ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, να χαιρετήσω καταρχήν και να καλωσορίσω τον Επίτροπο και να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την ενδελεχή ανάλυση που μας έδωσε στην κατάσταση για μια σειρά αποζητήματα. Δεν θα σταθώ φυσικά σε όλα αυτά τα θέματα και επομένως θα σας κουράσω. Θέλω απλώς να χαιρετήσω τα σχόλια του κ. Βητρόπου σε σχέση με το σύστημα PNR. Πάντα εγώ έχω συνεργαστεί με τους συναδέλφους μου προσπαθώντας να ικανοποιήσω τις επιθυμίες τους στην Επιτροπή μου Επιτροπή μας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός ότι η Κομισιόν θα φέρει τώρα νέες προτάσεις, νέες προ... προτάσεις τροποποιημένες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τις ανησυχίες των συναδέλφων, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και τις νέες αυτές προτάσεις. Θέλω να τώρα της Κομισιόν, θέλω να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο θυμίο. Θέλω να αντιμετωπίσουμε το θέμα των διαδικασιών και της επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένες εξελίσεις οι οποίες είναι αρνητικού χαρακτήρα και υπάρχει μεγάλη πίεση σε ορισμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει προσεκτικά τι διαφορέ και την ε, ε, ποικίλη ποιότητα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των αιτήσεων ασύλου και ιδίως τις διαφορές σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής των προσφύγων και κυρίως σε ό,τι αφορά τα παιδιά τους ανήλικους, κάτι το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα και την εκλογική μου περιφέρεια του εκλογής μου, είναι ότι ανεξάρτητα από τις ε, ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόσουμε στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, είναι απαραίτητο να έχουμε απόλυτη επίγνωση της ανάγκης να υπάρξει ένας ανθρωπιστικός τρόπος αντιμετώπισης των παιδιών. Επειδή λοιπόν ποικίλουν πάρα πολύ τα μέτρα σε επίπεδο ποιότητος και οι συνδίκες κράτησης των ανηλίκων και των παιδιών δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι ως Ευρωπαίοι, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ για την ομάδα Άλτε η Σεσίλια Βίξτρομ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο Αβραμόπουλο που ήλθε ενώπιον μας στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Έχω να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με τον κανονισμό του Δουβλίνου και τις ε, πρόνοιες σε σχέση με τους μη συνοδευόμενους ανηλίκους. Όπως ξέρετε στις διαπραγματεύσεις για τον νέο κανονισμό του Δουβλίνου αποφασίσαμε να επανέλθουμε και να επαξετάσουμε το άρθρο 8 για τους μη συνοδευόμενους ανηλίκους από τη στιγμή που θα υπήρχε μια απόφαση δικαστική για τις εκκρεμείς τότε υποθέσεις. Οι, τα τρία βασικά θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί να ευθυγραμμίσουν τον κανονισμό του Δουβλίνου με την δικαστική απόφαση, με τις δικαστικές αποφάσεις. Η Κομισιόν τήρησε το λόγο της και επανήλθε με μια πρόταση εφέτος το καλοκαίρι, κάτι το οποίο το εκτιμώ ιδιαίτερο. Η δική σας πρόταση ήταν ιδιαίτερα καλόδεκτη στην ΛΥΜΠΕ γιατί σέβεται την απόφαση των δικαστηρίων και επομένως σταματά την ε, άσκοπη μεταφορά ετούντων ασύλου από μία χώρα σε μία άλλη. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να ξέρω αν θα σταθείτε εξίσου στεναρός όπως ο προκάτοχός σας, προκάτοχός σας το να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και να μην αλλάξετε την πρόταση της Κομισιόν ώστε να κατέβει κάτω από το επίπεδο της απόφασης των δικαστηρίων. Γιατί τα δικαστήρια είπαν σαφώς ότι δεν πρέπει να μεταφέρονται από τη μία χώρα στην άλλη ως ένα εμπόρευμα, ως ένα πακέτο οι ανήλικοι. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν. Δεύτερον, θέλω να αναφέρω ότι για ορισμένους μπορεί να, μπορεί να έλθει και μία απόφαση για την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής ρύθμισης για το PNR. Αλλά ξέρετε ότι η Επιτροπή μας πριν από δύο χρόνια έχει απορρίψει αυτή την πρόταση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν κύριε Αβραμόπουλε, αν είσαστε επιγνώση του γεγονότος ότι το Ολλανδικό Κοινοβούλιο έχει απορρίψει την ιδέα ενός εθνικού συστήματος PNR και η κυβέρνηση των κάτω χωρών έχει σταματήσει το σχέδιο αυτό το οποίο χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρήματα θα επανέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τώρα τα εθνικά κοινοβούλια αντιτίθενται στα συστήματα PNR εθνικού χαρακτήρα, τι θα κάνετε. Θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε ένα υποχρεωτικό σύστημα PNR μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν γίνει κάτι τέτοιο και αν χρειάζεται προστασία δεδομένων και αυτό είναι μία από τις κύριες ανησυχίες μας γιατί εσείς μαζί με τους συναδέλφους σας στην Κομισιόν δεν αποδίδετε περισσότερη μέρημνα στον εξασφαλιστή ότι πρώτα θα εγκριθεί η οδηγία για την προστασία δεδομένων, γιατί αυτό θα είναι το κύριο, το κέριο ορόσημο το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να λειτουργούμε όταν αναλαμβάνουμε ε, μέτρα και ρυθμίσεις για την συλλογή δεδομένων. Αυτά ήταν λοιπόν δύο σημαντικά θέματα και νομίζω ότι τήρησε και το χρόνο μου. Προσβλέπω στο, στην απάντησή σας λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ Σίλια. Ο συντονιστής για την ΓΚΟΕ. Κορνίλια. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις, τα εισαγωγικά σας λόγια και την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της πολιτικής μετανάστευσης. Όταν εσείς μιλάτε για πολιτική μετανάστευση, υπάρχουν δύο ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε. Το πρώτο ερώτημα το οποίο θα ήθελα να ακούσω να απαντάτε είναι ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με το μέλλον του συστήματος ε, του Δουβλίνου. Έρχεστε από μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα λόγω του συστήματος αυτού. Έρχονται πάρα πολλοί ε, ετούντες άσυλο στη χώρα σας, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν, πιστεύετε, ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σύστημα, ε, θέλετε να επιμείνετε σε αυτό το σύστημα, να παραμείνει ως έχει ή θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις, βλέπετε την ανάγκη να υπάρξει αλλαγή σε αυτό το σύστημα. Ένα δεύτερο στοιχείο, όταν μιλάμε πάλι για μετανάστευση, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την επανεγκατάσταση των μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να προχωρήσει προ μια τέτοια ρύθμιση και τα κράτη-μέλη φυσικά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να ενισχύσετε την επανεγκατάσταση των μεταναστών και να πείσετε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν μαζί σα. Αυτά είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με το άσυλο και την μετανάστευση. Τώρα, εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ γιατί την προηγούμενη εβδομάδα πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η συμφωνία PNR μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά. Και είναι απόλυτα σαφές ότι μπορούμε να περιμένουμε μια ιδιαίτερα επικριτική απόφαση σε σχέση με τα στοιχεία αυτά της κράτησης ε, δεδομένων όταν δεν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι για αυτά. Και ξέρουμε ότι το PNR δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τέτοια μορφή κράτησης και ε, διατήρησης προσωπικών δεδομένων. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε τη στιγμή που έχει πάει αυτή η απόφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκκρεμεί δικαστική απόφαση, αν είμαστε σοβαροί όταν θέλουμε να κάνουμε μια συμφωνία τη στιγμή που εκκρεμεί η απόφαση στο δικαστήριο. Και μπορούμε να περιμένουμε μια αρνητική απόφαση ίσως. Μήπως θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν, μήπως αυτό είναι το ελάχιστο, να περιμένουμε τη δικαστική απόφαση και προσπαθούμε να τα κλείσουμε όλα αυτά πολύ γρήγορα, να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία. Μα τι θα γίνει αν αυτή η συμφωνία έρθει σε σύγκρουση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου, θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Τι θα κάνετε λοιπόν ώστε να εξασφαλίσετε ότι το πακέτο για την προστασία δεδομένων, το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό για μας, θα μπορέσει να εγκριθεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει πίεση ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί το πακέτο αυτό για την τα, προσωπικά δεδομένα και γι' αυτό πρέπει να αγωνιστείτε περισσότερο και όχι για το PNR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και η Σεσίλια και η Κορνίλια αναφέρθηκαν στην διατήρηση των δεδομένων, θα ήθελα και εγώ σαν Ολλανδέζα βουλευτής να ε, δώσω έμφαση στο θέμα αυτό και να πω ότι και εγώ ότι το κοινοβούλιο όμως είπε ε, όχι, δεν θα πάρουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για την νόμιμη μετανάστευση. Η Κομισιόν λέει ότι θα δημιουργήσει μια, θα προτείνει μια νέα πολιτική για τη μετανάστευση. Μα είπατε, Επίτροπε, ότι θέλετε να αλλάξετε την συζήτηση, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τη μετανάστευση. Και εγώ θέλω το ίδιο. Αλλά δεν καταλαβαίνω πόσο το να θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε για τη μετανάστευση όταν προσπαθούμε να βρούμε ε, ε, λειτουργικά ε, μέτρα για να καταπολεμήσουμε την, τους, τους όλους αυτούς τους ξένους πολεμιστές κτλ. και την καταπολέμηση την, των ακραίων ιδεολογιών και τρομοκρατικών ενεργειών κτλ. Πρέπει να σεβαστούμε τους ε, μετανάστες, ε, πρέπει να βρούμε τις, ποιες είναι οι νόμιμες μορφές μετανάστευσης. Και θα πρέπει, σύμφωνα με την άποψή μου, αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν στην, ε, Ευρώπη, που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, να, να μπορούν να ταξιδέψουν νόμιμα. Και υπάρχουν τρεις κατηγορίες ε, μεταναστών, αυτοί που ζητάνε άσυλο, αυτοί που, είναι, που έρχονται για για εργασία και δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες και αυτοί που διακινούνται ε, κρυφά δεν μπορούν να έρθουν νόμιμα στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να προτείνουμε νέες νέους νόμους, να υποβάλουμε νέες προτάσεις. Εσείς ε, περιορίσατε την πρόταση αυτή μονάχα στα άτομα τα οποία έχουν ε, ανώτερη εκπαίδευση. Και αυτό είναι περιορισμένο, διότι ούτω ή άλλω κάθε κράτο μέλο έχει τη δική του νομοθεσία για του ε, μορφωμένου, αν θέλετε. Θα πρέπει να δούμε την οδηγία για του ε, εποχιακά, εποχιακά αποσχολούμενου, για, τους, για το πώ θα μπορούσαμε να νομιμοποιήσουμε αυτού που αμείβονται με χαμηλούς μισθούς. Τότε και μόνο θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε την, μετανάστευση. Επίσης, η οι ΟΠΕΡ, αυτές οι γυναίκες που φροντίζουν και προσέχουν τα παιδιά. Αυτό έχει, δεν χρησιμοποιούνται σωστά, ε, δεν έχουν, ε, τους εκμεταλλευόμαστε, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αυτούς, για τα, για τα κράτη-μέλη συναντιόνται με χώρες της Αφρικής, ε, ε, συναντιόνται στην ε, Ρώμη και κάνουμε συμφωνίες με την Ερυθρέα για το πώς θα κρατήσουν τους μετανάστες στη χώρα τους, Νότιο Σουδάν και Ερυθρέα. Δεν νομίζω ότι συμβαίνουν κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, δεν ήθελα να σταματήσω μια και μιλούσαμε για την νόμιμη μετανάστευση. Ο τελευταίος συντονιστής η Λάουρα Φεράρα. Λάουρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Βραμόπουλα Και εγώ θα περιοριστώ, στην, θα εστιάσω την προσοχή μου στην νόμιμη μετανάστευση και θα συμφωνήσω με τα όσα είπε η κυρία Σαρτζεντίνη το να καταπολεμήσουμε την ε, παράνομη μετανάστευση και να εστιάσουμε την προσοχή μας στην νόμιμη μετανάστευση. Πάρα πολύ καλό αυτό. Ε, πολύ καλή και η οδηγία για τους ερευνητές και για τους φοιτητές, αλλά νομίζω ότι εξετάζουμε τον μετανάστη ε, από τη σκοπιά της ε, οικονομικής χρησιμότητάς τους και όχι σαν ανθρώπινο όν το οποίο απαιτεί να προστατευτούν τα δικαιώματά του. Το είπε η κυρία Σαρτζεντίνη, ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών έρχονται εδώ για να επιβιώσουν, γιατί θέλουν να ξεφύγουν από τις διώξεις, από τον πόλεμο και θα πρέπει ε, για τα άτομα αυτά να λάβουμε υπόψη μας ότι η οδηγία για την ε, Blue Card ή για την, ε, η οδηγία για τους ερευνητές και τους φοιτητές δεν αποτελεί μια απάντηση, μια λύση. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε νόμιμη πρόσβαση στην Ευρώπη. Ξεκινώντας από αυτό, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια ουσιαστική ε, προσπάθεια να καταπολεμήσουμε την ε, παράνομη διακίνηση των ανθρώπων. Όλοι θέλουμε να, καταπολε... να εξαφανίσουμε ε, τους διακινητές αλλά θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη νομοθετική βάση, πρέπει να έχουμε το σωστό νομικό πλαίσιο, γιατί θα πρέπει να λύσουμε εξάντε το, πρόβλημα προληπτικά και όχι εξπόστο. Επίσης η χρησιμοποίηση των πόρων. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί στην Ιταλία και πρόσφατα έγινε και μία έρευνα για το πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι για την μετανάστευση. Λοιπόν, στην Ιταλία η κατάσταση είναι απογοητευτική, ε, δεν, απο, δεν απορροφώνται τα χρήματα. Μία απόφαση του, του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου ε, λέει ότι στην Ιταλία δεν μπορούμε να επανενώσουμε μία οικογένεια διότι δεν εξασφαλίζεται η σωστή μεταχείρισή τους, η αξιοπρεπής ε, αντιμετώπιση τους και επηρεάζεται η όλη κατάσταση από την ε, αγκληματικότητα, από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κέντρα πρώτης ε, υποδοχής και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην σωστή χρησιμοποίηση των πόρων για τη μετανάστευση εν κατακλείδη τα, για τα θέματα της διαδικασίας ε, ταυτοποίησης ε, που επιτρέπουν στην Ιταλία και όχι μόνο εκεί να χρησιμοποιηθεί και ακόμα και η βία για να μπορέσει για να μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση, να, να βρεθεί δηλαδή η ταυτότητα των, ε, των ατόμων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων νομίζω ότι καλό θα ήταν να παρέμβετε και πάνω σε αυτό το θέμα. Uh, κύριε Επίτροπε, ε, τελείωσε ο γύρος ε, των συντονιστών, περνάμε στα μέλη και νομίζω ότι αφορά όλα, αφορούν όλα τα θέματα του χαρτοφυλακία τους, ήταν προβλέψιμο. Ε, τώρα σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από όλους άκουσα σχεδόν όλα εκείνα που σε ένα μεγάλο βαθμό κάλυψαν την αρχική μου εισήγηση σήμερα. Ωστόσο, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται σε κάποια σημεία να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω στην κυρία Μέτσολα ότι στο πρόγραμμα εργασίες του 2015 ε, θα δείτε την ε, Ευρωπαϊκή Ατζέντα επάνω στη μετανάστευση. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Χρειάζεται ολιστική προσέγγιση. Μελετώντας τους φακέλους μέσα από τα χρόνια που πέρασαν αφού του πρώτο εμφανίζεται σε αυτή τη νέα μορφή μετανάστευση στην Ευρώπη διεπίστωσα πρώτα απ' όλα ότι η Ευρώπη ευθυνδιάστηκε και στη συνέχεια άρχισε να ερμηνεύει διαφορετικά αυτό το φαινόμενο γιατί η μετανάστευση αυτής της περίοδου δεν έχει καμιά σχέση με τη μετανάστευση των περίοδων που προηγήθηκαν. Ακολουθήθηκε μια πολιτική, θα λέγα κατακαιρματισμένη, η οποία έφερε ωστόσο σε κάποιους τομείς αποτελέσματα. Σήμερα όμως βρισκόμαστε μπροστά σε μια εντελώς καινούργια πραγματικότητα. Και δεν κρύβω ότι προετοιμαζόμενος για την πρώτη μου εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής σας για την ακρόαση που έγινε πριν από 1,5 περίπου μήνα έμαθα και εγώ αν και προέρχομαι από την ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια πολλά από εκείνα που έχουν να κάνουν με αυτή τη νέα μορφή μετανάστευση. Και συμμερίζομαι απόλυτα με την Επιτροπή την ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνει στον ε, σεβασμό πάρα πολλά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σε καμία περίπτωση εγώ τουλάχιστον δεν θα επιτρέψω να διασυνδέεται το έγκλημα ή η τρομοκρατία με τη μετανάστευση. Είναι εντελώς διαφορετικά θέματα. Μόνο που η τύχη μου το θέλησε στο χαρτοφυλάκιό μου να έχω συγχρόνως και θέματα που αφορούν στην ασφάλεια της Ευρώπης και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ανάγκη να υιοθετηθεί, όπω είπα πρωτήτερα, απαντώ στο ερώτημά σα, μια ολιστική προσέγγιση του θέματο. Γι' αυτό είχα μιλήσει εξ αρχή ότι βασική στρατηγική κατεύθυνση τη νέα πολιτική για την μετανάστευση είναι να δημιουργηθούν οι όροι και οι προποθέσει για νόμιμη μετανάστευση. Και εκεί πάνω είναι που έδωσα πολλέ εξηγήσεις τι εννοούσαμε αυτό. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στην ανάγκη για συνεργασία. Αυτό έγινε στην Ρώμη προχτές. Σας το είπα και πριν. Στην Ρώμη για πρώτη φορά γύρω από το ίδιο τραπέζι κάθισαν χώρες προέλευσης, χώρες μέσω των οποίων διέρχεται το μεταναστευτικό ρεύμα, transit countries, και βεβαίω οι χώρες προορισμού. Και πρέπει να σας πω ότι φωτίστηκαν πολλές πτυχές από αυτήν την υπόθεση που σε πολλούς από εμάς δεν ήταν γνωστές. Δηλαδή, για πρώτη φορά συμμετείχαν και οι Αφρικανοί ε, εταίροι μας σε αυτή την προσπάθεια. Και θα δείτε ότι η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ σημαντική και χρήσιμη. Συμφωνείτε από ό,τι παρατήρησα για το ευρωπαϊκό PNR και βέβαια με παράλληλη ενίσχυση των data protection. Αυτή είναι η πολιτική μας. Το περιέγραψα με ιδιαίτερη σαφήνεια στην αρχή και το επαναλαμβάνω και τώρα. Σε ό,τι αφορά Τώρα αυτό που επεσήμανε η κυρία Ζήπερ. Γνωρίζω, τις απόψεις σας τις θυμάμαι και από παλιότερα, επιμένετε. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Πρέπει να συνεργαστούμε. Έχω μια άποψη, μια αντίληψη που να κάνει με την κοινοβουλευτική διαδικασία. Εμείς ως Commission, ε, αν θέλετε ως κυβέρνηση της Ευρώπης, ελεγχόμεθα από το Κοινοβούλιο. Αλλά ζητούμε και από το Κοινοβούλιο να συνεργάζεται μαζί μας. Γιατί το τελικό συνθετικό αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στο να αφήσουμε πίσω μας μια πολιτική κληρονομιά με μέτρα, αποφάσεις, νομοθεσίες που θα έχουν συμβάλει συνολικά στο να έχει κινηθεί η Ευρώπη προς τα εμπρός. Εγώ αυτό ήθελα να σας δείσω. Βεβαίω με πλήρη σεβασμό των απόψεων που διατυπώνονται. Γνωρίζω και τις επιμέρους ευαισθησίες ή και τις σταθερές ιδεολογικές απόψεις που στηρίζονται σε αρχές και αξίες και τις σέβομαι ιδιαίτερα. Έδωσα λοιπόν με σαφήνεια πιστεύω το στίγμα της πολιτικής που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Απόλυτη προστασία από τη μία πλευρά των θεμελιωδών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη μεριά μια πιο δυναμική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Γιατί υπάρχει κανείς σε την αίθουσα που διαφωνεί ότι η τρομοκρατία είναι μια πραγματικότητα. Ότι καθημερινά αγωνιούμε, κοιμόμαστε με την αγωνία τι θα συμβεί την επόμενη μέρα μετά όσα γίνονται στον ευρύτερο γεωπολιτικό μας χώρο με ό,τι αυτό συνοδεύει ανεξέλεγκτες τρομοκρατικές δραστηριότητε δεν πρέπει εκεί η Ευρώπη να ορθώσει το αναστημά Δεν πρέπει την ίδια στιγμή να αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα όχι μόνο αυτό το φαινόμενο, αλλά και ό,τι διασυνδέεται με την ε, μετανάστευση και αναφέρομαι στους μάγκλες και τους τράφικες, Δεν πρέπει εκεί οι ποινές να είναι πάρα πολύ αυστηρές. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα επιχειρησιακού τύπου επέμβασης. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις άλλες χώρες. Ήδη αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πώς αυτή η βιομηχανία έχει στηθεί. Και πρέπει να σας πω κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί και να σας εκπλήξει. Αλλά πολλές από αυτές τις οργανώσεις είναι καλύτερα εξοπλισμένες ακόμα και από τα ίδια τα κράτη. Έχουν στη διάθεσή τους πολύ προηγμένες τεχνολογίες. Και δοκιμάστηκε αυτό στην πράξη στη συλλογική προσπάθεια που όλοι καταβάλουμε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παράνομης αυτής εγκληματικής διακίνησης ανθρώπινων ψυχών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Έθιξε ο κύριος Κύρκο και τον ευχαριστώ ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Commissioner, before you um, get on to Mr. Kirkhope, may I just respectfully um, mention that when you finish with the commissioners, we have 25 members who will be asking questions, all deserving of an answer. So I just wanted to put that figure into your subconscious. So um, it's certainly in mine. Um, so just speed up a Έχουμε πολλά μέλη που θα θέλουν να λάβουν το λόγο. Οπότε, αν θέλετε να επιταχύνετε λιγάκι, γιατί υπάρχουν και 25 μέλη τα οποία θέλουν να θέσουν ερωτήματα και δεν θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Αν μπορείτε λοιπόν να επιταχύνετε λίγα με τους συντονιστές. Ε, within maybe within the conscious, my, my conscious <laughs> response to my unconscious reactions. Λοιπόν, υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της ε, συνειδητής μου ε, απάντησης και αυτών που θέλω υποσυνείδητα να πω. Uh, members are conscious that you can't answer everything speedily and you will be back. So I think call... Θα έχετε την ευκαιρία να επανέλθετε, λέει ο, ο κύριος Μωράης, οι συνάδελφοι ξέρουν ότι θα επανέλθετε λοιπόν να μην σα απασχολεί το θέμα αυτό. Ήθελα επίση να πω στην κυρία Μέτσολα για την ηθαγένεια της ε, Μάλτα. Να μην λησμονούμε ότι αυτό είναι καθαρά εθνικό θέμα. Όμω, όσον αφορά στι επιπτώσει που ίσω είχε και στην ευρωπαϊκή ηθαγένεια θα το δούμε με την ε, ε, Επίτροπο κυρία Ζούροβα η οποία έχει και την αρμοδιότητα. Άρχισα πριν από λίγο λοιπόν να απαντώ και να πω στον κύριο Κυρκόπον ότι προφανώ χρειάζονται βελτιώσει στο σύστημα ασύλου και η Επιτροπή το παρακολουθεί. Όσον αφορά τώρα στο PNR, όντως θέλουμε ε, μαζί σας κύριε Συγητά να δουλέψουμε. Οι βελτιώσεις όλων των σημείων που, θίγεται, που θίγονται σήμερα θα γίνουν μαζί με εσάς. Ε, η, η Επιτροπή, πρέπει να σας πω κυρία Βίξτον, δεν έχει σκοπό να χαμηλώσει τα στάνταρτς δεν πρόκειται να κάνει καμία παραχώρηση στις βασικές θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται αυτή η πολιτική. Ξέρω πράγματι ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ απέρριψε το ε, Ευρωπαϊκό PNR, το EU Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το βελτιώσουμε. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για την Ολλανδία, πρέπει να σας πω, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι στην Επιτροπή έχουμε σταθμίσει με ιδιαίτερη προσοχή ε, τις καταστάσεις πριν ε, σας παρουσιάσουμε την, ε, την πολιτική μας. Ε, δεν θα ήθελα να πάρω παραπάνω χρόνο τώρα γιατί ξέρω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ερωτήσεις αλλά θα ήθελα απλώς να πω ότι μια παρατήρηση ότι το PNR είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το data retention. θα ήθελα να σας καλέσω, το είπα και στα εισαγωγικά μου, σε μια πιο ρεαλιστική συνεργασία σταθμίζοντας, όπως είπα, όλες τις ε, εναλλακτικές. Ε, όσον αφορά στο data retention, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να κινηθώ με βιασύνη. Εκκρεμούν και οι αποφάσεις των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων, τις οποίες περιμένουμε. Θα επανέλθουμε με οδηγό βεβαίω την απόφαση του δικαστηρίου. Τέλος για την κυρία Σαρτζετίνη θα ήθελα να πω ότι και το δεν έκανε καμία σύνδεση Τις τρομοκρατίες και των foreign fighters με τους ε, μετανάστες. Αναφέρθηκα συνοπτικά σε τομείς ε, του χαρτοφυλακίου και της πολιτικής μας. Και βέβαια κλείνω λέγοντας ότι η νόμιμη μετανάστευση είναι ο μόνος δρόμος και πάνω σε αυτή δουλεύουμε για να παρουσιάσουμε σύντομα θέλω να πιστεύω και μέσα στο προσεχές εξάμεινο μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση μιας νέας χάρτας για τη μετανάστευση. was Laura uh, uh, But there was there was um, Laura Ferrara. oh. Did you mention? Also in legal migration. Yes. Αναφέρθηκα πριν στην ε, νόμιμη μετανάστευση. Αυτό εννοούσε προφανώς και η κυρία Φεράρα. Και το επαναβεβαίωσα και στην αρχή της απαντησής μου και τώρα. Okay, um, θα περάσουμε στα μέλη. Έχουμε 25 μέλη. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Είχα ε, ένα, ένα ερώτημα ε, συγκεκριμένο στη συμφωνία του Δουβλίνου για τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Σε καμία περίπτωση σας αναφερθήκα ότι όταν είπα ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αλλάξουμε γραμμή από αυτή που γνωρίζετε και που έχουμε θέσει. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος. Okay. Απλώς και εγώ ήθελα να πάρω μία απάντηση. Απάντηση σε αυτά τα οποία είπα όσον αφορά τους νόμους, τρόπους ε, διακίνησης, ε, μεταφοράς ε, τρόπους ε, προσέγγισης κτλ. In fact... Οι νόμιμοι δρόμοι και τα προβλήματα με, το, με την ταυτοποίηση. είναι τα θέματα της, του, του, του τρόπου με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε την μετανάστευση, τα όσα λέμε για τη μετανάστευση. Ναι, μίλησε για τους νόμιμους δρόμους ο Επίτροπος. Μπορώ να σας το ε, διαβεβαιώσω και εγώ, αλλά ήταν μέσα στην ζέση του πολέμου, αν θέλετε. Κορνίλια, Κορνίλια. Είναι διαδικαστικό το θέμα. Πες τι θέλεις να πεις. Κοιτάξτε, είμαι ένα υπομονετικό άτομο γενικά, αλλά ούτε μία από τις ερωτήσεις μου δεν έτυχε απάντησης. Θα ήθελα να έχω μια απάντηση από εσά. Πιστεύετε ότι τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό PNR παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα η συμφωνία PNR με τον Καναδά έχει έλθει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η οδηγία για την κράτηση δεδομένων δεν ισχύει. Να συνεχίσουμε ε, στην κατεύθυνση αυτή και δεν... Μα ήμουν σαφής όπως με ειλικρίνεια θέτε τις ερωτήσεις σας, με ειλικρίνεια σας απαντώ και εγώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε για την, ε, στην ίδια γραμμή, δηλαδή για ένα ευρωπαϊκό ε, ε, PNR. Σε ό,τι αφορά την, το αίτημα για μια νομική γνώμη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε ό,τι αφορά το EU Canada PNR, εκεί περιμένουμε να δούμε. Νομίζω στα εισαγωγικά ήμουν απόλυτα σαφής σε αυτό το σημείο. Όχι, όχι, όχι, φτάνει. Τώρα θέλουμε πειθαρχία. Έχουμε 25 μέλη που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις και ε, πολλοί θα είναι εισηγητές, υπήρξαν εισηγητές ε, και θα πρέπει να, να θέσουν ερωτήσεις και να πάρουν απαντήσεις, διότι είναι αδικό για αυτούς στην πρώτη συνάντηση με τον Επίτροπο. Λοιπόν, δεν θέλουμε να συνεχίσετε με τις ερωτήσεις σας δύο λεπτά και σας παρακαλώ πειθαρχία να τηρείτε το χρόνο σας. Αν θέλετε και λιγότερο από δύο λεπτά θα ήταν καλύτερο. Θα επανέλθει βεβαίω ο Επίτροπος όπως το υποσχέθηκε. Κυρία Κυρία Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ για την εισήγησή σας. Ε, θα αναφερθώ στις συμφωνίες επανεισδοχής της ευρωπαϊκής ένωσης με τρίτες χώρες που κι εσείς έχετε επισημάνει ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο κατά της παράνομης μετανάστευσης από το δεδομένο ότι εγγυώνται τις καλές σχέσεις και τη συνεργασία της ευρωπαϊκής ένωσης με τις χώρες αυτές από τη μια πλευρά και από την άλλη δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα σε εκείνους τους διακινητές τους εγκληματικών πράξεων που διακινούν ανθρώπους και εμπορεύονται ανθρώπους. θέλω να σας ρωτήσω επειδή με το δεδομένο ότι αυτές οι συμφωνίες με τρίτες χώρες τελευταία, ε, τα τελευταία χρόνια έχουν διευρυνθεί αν προβλέπετε μια περαιτέρω διεύρυνση τέτοιων συμφωνιών και επίσης ε, να σας ρωτήσω εάν ε, ε, έχει μελετηθεί από την επιτροπή η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των συμφωνιών αυτών. και μια δεύτερη ερώτηση παρακαλώ έχουμε σαν δεδομένο ότι υπάρχουν τρίτες χώρες που παρά το γεγονός ότι έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες δεν τις στηρούν και δεν τις σέβονται. ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος πιεστικός μοχλός αλλά ίσως να υπάρχουν στην επιτροπή σκέψεις για μια λύση έκτακτης ανάγκης για μια άλλη στρατηγική που μπορεί να ακολουθηθεί σε αυτή την κατεύθυνση το δεδομένο ότι όλοι συμφωνούμε ότι επαναλαμβάνω είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην κατεύθυνση της νόμιμης μετανάστευσης που περιλαμβάνεται ως κυρίαρχο θέμα και στην ατζέντα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τηρήσατε ε, τον χρόνο Άννη Γκόμες. Κύριε Πίτροπε, βεβαίως όσα είπε η Τζούντιθ Αντζεντίνη συμφωνώ ότι Έχουμε το Σουδάν, την Ερυθρέα, την Αιθιοπία. Αυτές τις κυβερνήσεις υπάρχει, ε, υπάρχει πόλεμος εναντίον ανθρώπων και γι' αυτό φεύγουν από τη χώρα τους. Ε, συμφωνίες με αυτές τις χώρες. Αρχίσατε να μιλάτε για τους μετανάστες που βάζουν τη ζωή τους στα χέρια των ε, λαθροδιακινητών ε, και δεν υπάρχουν νόμιμοι οδοί για αυτούς τους μετανάστες. Αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσω για μερικούς μετανάστες στους οποίους τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι, όχι μόνο ε, δίνουν πράσινη κάρτα αλλά στρώνουν και το κόκκινο χαλί δεν είναι ένα θέμα τελείως εθνικό, είναι θέμα ευρωπαϊκό. Ε, είναι η ακαιρεότητα του συστήματος Schengen που διακυβεύεται και η δική μας ακαιρεότητα, διότι είναι ένα σύστημα εισαγωγής οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς. Και μιλάω για τη χώρα μου και δεν είναι η μόνη Πορτογαλία, ξέρετε πριν μερικές εβδομάδες, ο επικεφαλής αστυνομία αστυνομίας συνελήφθη, επίσης ένα αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Μητρών, σε ένα δίκτυο ε, αξιωματούχων της δίκησης, διότι ήσαν σε ένα δίκτυο που ε, εκμεταλλευόταν τις θεωρήσεις δεν είναι μόνο ευκαιρίες για διαφθορά, είναι το σύστημα το ίδιο. Δεν έχει τους ελέγχους που χρειάζονται, κυρίως για το ξέπλυμα χρήματο. Ο Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας είπε ότι ε, για τους ελέγχους ρώτησα τον Υπουργό και δεν έλαβα απάντηση. Ήθελα ονόματα, ονόματα άνω των 3.000 ατόμων που έλαβαν χρυσές θεωρήσεις ε, στην Πορτογαλία, διότι δεν είναι μόνο συγγενείς, ε, χρησιμοποιώντας ε, την προστασία δεδομένων δεν έλαβα απαντήσεις. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Δεν είναι μόνο ανήθικο, είναι ε, κατά το, της αρχής ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που δεν μπορεί να συνεχίσει να παραβλέπει η Κομισιό. Συσπινότα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Στον έκτη έκθεση για την λειτουργία της χώρου Σέγγεν που μας παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί γίνεται λόγος σαφώς ότι παρόλο που το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να αποφανθεί για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με τη Βουλγαρία και την Ρουμανία, η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρω την προσχώρηση Βουλγαρίας και Ρουμανίας στον χώρο Σέγγεν. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη δέσμευση Τη της Επιτροπής, ποια είναι τα επόμενα στάδια και τα μέτρα, ούτως ώστε να προσχωρήσει η Βουλγαρία και η Ρουμανία στον χώρο Σέγγεν και αυτό να γίνει πραγματικότητα σε προσεχές μέλλον. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις διευκρινήσεις που θα μας δώσετε για αυτήν την συγκεκριμένη διαδικασία για την πλήρη συμμετοχή των δύο αυτών χώρων στο ευρωπαϊκό αυτό σχέδιο και το οποίο οι δύο χώρες περιμένουν εδώ και καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Επίτροπε. Στην ακρόαση ή μας είπατε ότι θέλετε να υπάρχει ένα κοινό σύστημα ασύλου. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε εσείς αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα. Εδώ και μία εβδομάδα είναι γύρω στους 200, 200 Σύριοι οι οποίοι κάνουν απεργία πίνης πίνας στο, στην πλατεία συντάγματος. Παιδιά, άτομα τα οποία τα πήγαν στο νοσοκομείο. Είναι μία κατάσταση περίεργη. Θέλουν να προχωρήσουν προς μία τρίτη χώρα, αλλά είναι μπλοκαρισμένοι στην χώρα άφηξης σύμφωνα με τη συμφωνία του Δουβλίνου η κυβέρνηση δυστυχώς δεν μπορεί να χορηγήσει άσυλο, ούτε εργασία όμως. Έχουμε επομένες ζώνες όπου απουσιάζει το δίκαιο και υπάρχουν, υπάρχουν χώρες ε, τελικά όπου δεν, δεν μπορεί να γίνουν σεβαστές οι, οι διατάξεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπε και η κυρία Φεράρα, το δικαστήριο του Στρασβούργου δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις ε, κατάλληλες ε, συνθήκες υποδοχής. Επομένως, διαρωτώ με τι μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση στην Ελλάδα και μήπως ε, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να περιμένουμε μια μαζική ροή, ένα μαζικό ρεύμα μεταναστών που θα απαιτούσε την τροποποίηση της οδηγίας του 2001 όσον αφορά την αλληλεγγύη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μήπως θεωρείτε ότι θα έπρεπε να επανεξετάσουμε τον κανονισμό του Δουβλίνου 3 για να μην δημιουργούνται αυτές οι παράλογες καταστάσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε σε μια τρίτη χώρα οι μετανάστες και η χώρα υποδοχής δεν μπορεί να τους κρατήσει. Ευχαριστώ. Κυρία Σας Κύριε Πρόεδρε. Η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μας έδωσε λεπτομερείς εκθέσεις για την κατάσταση των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα χερσαία και στα αεροδρόμια. Η μεταρρύθμιση του κανονισμού και του 2001 και η στρατηγική του, της υπηρεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν βελτιώσει την κατάσταση. Η Frontex παραμένει πάντα σε ένα επίπεδο αδιαφάνειας και μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Η Έμιλι Οράιλι, η της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε να υπάρξει ένας μηχανισμός ατομικών προσφυγών σε περίπτωση δράσεων της Frontex έναντι μεταναστών. Θα μπορούσε η Κομισιόν να δεχτεί να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα. Ευχαριστώ. Uh, Κυρία Χολμάια. <laughs> komme gerade aus den Haushaltsverhandlungen, da gibt es auch etwas schwierige Kosten. Έρχομαι από κάτι διαπραγματεύσεις όπου υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σα. Ελπίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά και δύσκολα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα το ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με την ε, κατάσταση της Μεσογείου πώς θα αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι από τη μια μεριά έχουμε πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν καμιά ελπίδα να ζήσουν στη χώρα τους, να παραμείνουν στη χώρα τους και δεν έχουν φυσικά και καθόλου νόμιμους τρόπους μετανάστευσης στην Ευρώπη. Από την άλλη μεριά πώς θα αντιμετωπίσουμε τους διακινητές οι οποίοι με εγκληματικό τρόπο εκμεταλλεύονται την απόγνωση αυτών των ανθρώπων, πώς θα εμποδίσουμε λοιπόν την ε, διατήρηση των δικτύων αυτών διακίνησης. Και έχουμε επίσης και το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της, που έχει δυσχερανθεί πάρα πολύ λόγω της ε, τρομοκρατικής δράσης του Ισλαμικού κράτους και της απόλυτης ε, έλλειψης οποια, της ασυνειδησίας με την οποία έχει δράσει. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να εμποδίσει τους ξένους μαχητές να δρούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουν σε τρομοκρατικές ενέργειες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι εδώ μέσα στην Ευρώπη οι νέοι θα προσιλητίζονται από αυτές τις απόλυτα παράλογες και λανθασμένες ιδέες και θα προσελκύονται στην τρομοκρατία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό. Φυσικά έχετε πάρα πολλά θέματα όπως έχουμε και εμείς για τα ζητήματα αυτά. Thank you for sticking to time. Ευχαριστώ Μόνικα. Ο κύριος Κύρκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας βλέπω. Ε, να προσθέσω και εγώ για την κυρία σε αυτό που είπε η κυρία Σπινέλη, ε, οι πρόσφυγες στην Ελλάδα που κάνουν απεργία δεν θέλουν να κάνουν αίτηση για άσυλο θέλουν να του δοθούν χαρτιά ταξιδιωτικά για τι υπόλοιπε χώρε. Ένα ζήτημα που αφορά την επανεγκατάσταση. Μήπω θα μπορούσε και στη συνάντηση που έχετε τη Δευτέρα για αυτά τα θέματα να τεθεί ειδικά για του Σύρου πρόσφυγες που είναι μια περίπτωση ανθρώπων που σίγουρα θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, οι δυνατότητες επανεγκατάστασης να γίνει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα αποδεκτή. Η κοινωνική κυβέρνηση ξέρω πως δεν μπορεί να τους δώσει σαν τα χαρτιά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν και από τη σειρά τους να πεθάνουν από το κρύο και την πείνα στην πλατεία συντάγματος. Και το δεύτερο είναι, ε, την 1η του Γενάρη 600 παιδιά στην Ελλάδα θα μείνουν έξω από μη κυβερνητικέ οργανώσει που τα φιλοξενούν. Γίνεται αναδιάρθρωση των ταμείων τη μετανάστευση και, ε, και υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό. Έχει καθυστερήσει πολύ, κάτι πρέπει να γίνει γιατί οι οργανώσει μπορούν να καθυστερούν τι πληρωμέ του αν ξέρουν ότι έρχονται χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν από πού θα τα πάρουν. Οπότε θα έπρεπε ή δυνατόν κάτι να γίνει. Είναι 600 παιδιά και με και άλλε χώρε τη Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερη αριθμή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Kirkos. And we're, we're now obviously Getting. Κύριε Επίτροπε, ε, ακούμε και άλλα θέματα πέραν του, του, κυρίου θέματος που μας απασχολεί. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσάς, όχι μονάχα τους συναδέλφους, ε, ε, θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές, γιατί υπάρχουν και άλλα 12-13 μέλη που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ή θέλετε να ακούσετε όλες τις ερωτήσεις και να απαντήσετε μετά. Να είμαι ειλικρινής, προτιμώ να απαντήσω τώρα σε αυτές τις ερωτήσεις. Επομένως, συμφωνείτε κι εσείς ε, τα, τα μέλη της Επιτροπής μας ε, να ακούσουμε μια πρώτη δόση απαντήσεων από πλευρά του Επιτρόπου και μετά να ακούσουμε το δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να πω στην κυρία που έβαλε την πρώτη ερώτηση ότι ναι, προωθούμε τις διεθνείς συνεργασίες, δουλεύουμε αυτόν τον καιρό με περισσότερες χώρες από ό,τι συνεργαζόμαστε ε, πριν ε, και βέβαια προωθούμε όλα αυτά τα mobility partnership agreements τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία στα χέρια μας. Η φύση των συμφωνιών αυτών είναι, είναι πολυμερής ε, θα έλεγα ε, και βέβαια αναφέρομαι στην ελεύθερη, ε, στη free visa και στην ε, επιστροφή. Άρα είναι πολύ σωστό αυτό που επισημάνατε με την, με την ερώτησή σας. Εξάλλου πριν από λίγο αναφέρθηκα με σαφήνεια στο σημείο αυτό που θίξατε. κυρία Γκομέζ, πιστεύω στο διάλογο ε, sorry but I'm addressing to you right now εγώ μας πιστεύω στο διάλογο, όπως πιστεύετε και εσείς. Ε, μαζί με συναδέλφους επιτρόπους, διότι πρέπει να σας πω ότι στα πλαίσια της Κομισιόν υπάρχουν συνέργειες αυτόν τον καιρό όσον ε, τα θέματα και οι αρμοδιότητες ε, διασταυρώνονται, έτσι ώστε να μην υπάρξει από καμία πλευρά κανένα κενό στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε. Συζητούμε λοιπόν όλα τα θέματα πολιτικής ε, ανάπτυξης, με αντίστοιχα ωφέλη για την βελτίωση την οποία βλέπουμε των επιπέδων ε, θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων τόσο με τον κύριο Τίμερμανς όσο και με την κυρία ε, και έτσι αυτόν τον δρόμο ακολουθώντας πιστεύω ότι και οι πολιτικές που γερτούνται στο τέλος ε, θα διαμορφώσουν ένα σύστημα σταθερών μέσα στο, στην, στους κόπους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναφορικά τώρα με την Ρουμανία και την Βουλγαρία. Το είχα πει και στην την περίοδο, μάλλον την εποχή που προετοιμαζόμουν και απήντησα σε εσά στην ακρόαση που έγινε. Είναι ξεκάθαρο. Βεβαίως και η Επιτροπή μένει σταθερή στην απόφαση που έχει πάρει για να ανοίξει, ανοίξουν οι πόρτες της Σέγγεν και για τη Ρουμανία και για την ε, Βουλγαρία. Πιστεύουμε ότι με την προσαρμογή των δύο αυτών χωρών στους βασικούς όρους λειτουργίας της ζώνης Σέγγεν και με την βοήθεια που παρέχει ήδη η Επιτροπή τόσο στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, το σύστημα και εκεί θα λειτουργεί αποτελεσματικά. Είναι αλήθεια ότι έχουν ακουστεί και διαφορετικές ε, απόψεις, όπως είναι αρκετοί εκείνοι που αμφισβητούν την δυνατότητα των δύο αυτών ευρωπαϊκών χωρών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η Επιτροπή όμως θα του βοηθήσει, θα τι βοηθήσει και θα συμπαρασταθεί στην προσπάθεια που καταβάλουν αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσει των δύο χωρών και με βέβαιο ότι σύντομα και η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα είναι μέλη τη ζώνη Σέγγεν. Ε, αναφέρθηκε η κυρία Σπινέλη αλλά και ο κύριο ε, Κύρκο σε αυτό που πράγματι υπάρχει, ε, υπάρχει από τον καιρό στην Αθήνα. Θα ήθελα να σας πω ότι ήδη εγώ ενημερώθηκα από τις ελληνικές αρχές. Μάλιστα πρόσφατα βρέθηκα κάτω για μια γενικότερη συζήτηση και είμαι σε θέση να γνωρίζω πώς έχει κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, ε, αυτή η ομάδα Σύριων προσφύγων δεν ε, δέχεται, ενώ το προτείνει η ελληνική πλευρά, να υποβάλει ε, αίτημα για την χορήγηση ασύλου. Και τους λόγους τους γνωρίζετε. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι εκεί υπάρχει ένα κενό. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι είμαι σε θέση πάλι να γνωρίζω, οι ελληνικές αρχές ε, προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια σε αυτή τη φάση στους ε, ε, ε, Σύριους που βρίσκονται ε, συγκεντρωμένοι στην πλατεία συντάγματος στην Αθήνα. Την Δευτέρα, όπως ξέρετε και σας το είπα και πριν, θα μεταβώ στη Γενέβη όπου θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα αυτό, δηλαδή των Σύριων προσφύγων, που αυτό τον καιρό το ρεύμα αυξάνει όλο και περισσότερο γιατί η πίεση που ασκείται σε αυτό το λαό είναι ε, ιδιαίτερα πιεστική αυτή την περίοδο. Ε, αυτό που λέμε όμως για την Ελλάδα δεν ισχύει μόνο η ισχύει για όλες τις χώρες. Η απόφαση για το αν τελικά θα ζητήσει κάποιο άσυλο, όπως γνωρίζετε, είναι μια προσωπική επιλογή του ενδιαφερμένου και δεν υπάρχουν, εδώ έχουμε ένα κενό, νομικές δυνατότητες για ένα κράτος μέλος να πείσουν ένα πρόσωπο να το κάνει. Έστω και αν οι ανάγκες προστασίας αυτού του προσώπου είναι προφανής. Ωστόσο, <clears throat> θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι εδώ, ότι τα κράτη-μέλη έχουν την νομική υποχρέωση να ταυτοποιούν και να καταχωρούν τα πρόσωπα αυτά σωστά, ανάμεσα στα άλλα ε, και βεβαίως με την ε, λήψη ε, των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων. Δεν το δέχονται. Αυτό παρατηρείται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Όσον αφορά τώρα ε, για, τους, για Σύριους υπάρχει, υπάρχει συνένεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη ότι καμία επιστροφή εθελοντική ή καταναγκαστική δεν θα συντελείται λόγω της κατάστασης στη Συρία ανεξάρτητα από, την, από τη φύση της παραμονής των προσώπων αυτών στο έδαφος ε, του εν λόγω κράτους ε, μέλους. Και η Ελλάδα, όπω ξέρετε, δεν μιλάω σαν Έλληνα αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι σε θέση να το γνωρίζω γιατί με ενημέρωσαν οι ελληνικέ αρχέ. Εφαρμόζει ήδη από το 2010 ένα πρόγραμμα ασύλου για τη διαχείριση τη ε, ε, μετανάστευση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συστημικέ ελλείψεις που έχουν παρατηρηθεί και έχουν καταγραφεί. Εμεί τώρα, ω Επιτροπή από την άλλη πλευρά, ήδη όπω είπα και στην αρχή, έχουμε αναλάβει ε, μια πρωτοβουλία. Θα το συζητήσω και ε, με τους συναδέλφους τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά μεθαύριο θα είναι ένα από τα θέματα που θα θίξουμε σε ε, διεθνές πλέον επίπεδο ε, στην Γενέβη. Όσον αφορά τώρα την Frontex και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ναι, επιμένουμε σε αυτόν. Κάθε αναφορά που γίνεται και υπάρχουν πολλές θα ερευνάτε. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς η Κομισιόν αλλά και εσεί ασκείτε έλεγχο και οι πληροφορίε που κατά καιρού έρχονται μέσω του Κοινοβουλίου ελέγχονται από την Επιτροπή. Okay, we, we need to, we need to really... Τώρα θα πρέπει να επιτεχύνουμε την όλη διαδικασία. Διαδικαστικό. Κύριε Επίτροπε, τι είδους υποστήριξη, τι είδους υποστήριξη προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν τροφή, δεν υπάρχει τροφή. Τα άτομα πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Εσείς από πού βρήκατε τις πληροφορίες αυτές. Το, μα εσείς μου το είπατε πριν ότι πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν είναι μια παροχή βοήθειας. Από ό,τι πληροφορούμε ε, ήδη διατίθενται και τρόφιμα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι κάνουν αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι στο δρόμο συμφωνώ μαζί σας αυτό που λέτε. Εδώ υπάρχει ένα κενό, σας το περιέγραψα πριν. Αλλά η εικόνα που έχω είναι η εικόνα που μου δίνουν οι αναφορές που έρχονται από την Αθήνα. Αν έχετε κάποια διαφορετική, ευχαρίστω να σας ακούσω και να το ελέγξω. Okay. Thank you, Commissioner. Let's, let's move on to Mrs. Ας περάσουμε στην κυρία Μέιερ, που είναι η επόμενη ε, ομιλήτρια. Ehm, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω στον Επίτροπο. Προτίθεται ο Επίτροπος ε, να δημιουργήσει κέντρα υποδοχής σε αφρικανικές χώρες. Μήπως αυτό θα έλυνε κάπως, θα έδινε μια λύση στα, ε, στην κατάσταση. Επίσης με με βάση πρόσφατες δημοσιεύσεις στον τύπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να δημιουργήσει ένα ε, πανευρωπαϊκό σύστημα ε, ελέγχου των συνόρων. Τρίτον, για τους ε, πολεμιστές της τζιχάντ, για τους τζιχαντιστές, που υποτίθεται ότι επιτρέπεται να φύγουν αλλά δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν. Έχουμε ε, στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στον τύπο για τσιχαντιστές οι οποίοι εγκαταλείπουν την Ευρώπη και ποσοστό αυτών που επιστρέφει. Εσείς γνωρίζετε συγκεκριμένα στοιχεία πόσοι φύγανε και πόσοι επέστρεψαν. Ευχαριστώ, Κλοντ. Επειδή δεν έχουμε και χρόνο και λόγω των περιστάσεων, δεν έχω ερωτήσεις να κάνω. Απλώς κάποιες προτάσεις ή κάποιες ενθαρρύνσεις Καταρχάς για το PNR. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, να δημιουργήσουμε αυτό το ευρωπαϊκό PNR. Και αυτό απλώς και μόνο για να είμαστε και σε θέση ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα με τις άλλες ε, χώρες του πλανήτη που έχουν ε, σύστημα PNR. Επομένως δεν βλέπω για ποιο λόγο θα έπρεπε τώρα να σταματήσουμε την προσπάθεια να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας στον τομέα αυτό. Τώρα, κάτι άλλο τελείως διαφορετικό, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια ήπειρο, η οποία με, ενδιαφέρε, με ενδιαφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, την Αφρική. Ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε ε, με την Αφρική, έτσι ώστε να ελαφρύνουμε κάπως ε, την κατάσταση για τους μετανάστες ε, που έρχονται με διάφορα επίπεδα θέλησής τους. Ξέρω ότι για την Αριθρέα υπάρχουν πάρα πολλοί που θα ήθελαν να μείνουν στην Ερυθρέα. Όμως η Ερυθρέα έχει γίνει μια ανοιχτή φυλακή και για, και για αυτή τη χώρα θα πρέπει να ε, ε, υιοθετήσουμε μια διαφορετική ε, πολιτική. Η ενίσχυση των κρατών στην Αφρική. ξέρω ότι δεν, είναι, δεν είσαστε εσείς το δικό σας χαρτοφυλάκιο που είναι υπεύθυνο. Όμως, εσείς αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε είναι ότι εάν ε, δεν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κράτη σταθερά στο, στην νότια ακτή της ε, Μεσογείου, τότε η μετανάστευση θα, η κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση θα επιδεινωθεί και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ Φρανκ ο Χουάν Φερνάντο Αγγιλάρ, Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ για λόγω έλλειψης ε, του χρόνου. Θα, είμαι... θα, σας... θα στείλω ένα τηλεγράφημα. Έχω πολλές ερωτήσεις βέβαια που αφορούν ε, το συνδυασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και συνοριακών ελέγχων για τις ε, θεωρήσεις, για την υποχρεωτική εκπροσώπηση που είναι η πρόθεσή σας ε, να είσαστε, ε, θέλετε να το στείλετε ένα συγκεκριμένο μήνυμα για το τι θα γίνει εδώ, για τις επιστροφές δεύτερο. Είχαμε μια συζήτηση στην Ολομέλεια του Στρασβούργου την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρω ότι θα πρέπει να δοθεί μια συνέχεια καλό θα είναι να ακούσουμε περαιτέρω πληροφορίες. Τρίτο ερώτημα, ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, αλλά τώρα είναι η δική σας ε, σειρά. Τέταρτο θέμα την έκθεση που ακούσαμε σήμερα το πρωί από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για, τις, ε, για την κατάχρηση και την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα αεροδρόμια αλλά και στα ε, χερσαία σύνορα. Τι θα κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και ε, τελικά ένα σχόλιο. Υπάρχει μία απόφαση του, σχετικού, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα δικαιώματα των LGBT. Ε, άτομα τα οποία είναι υποχρεωμένα ας πούμε στις κάτω χώρες, ε, στους ελέγχους των συνόρων, να δηλώνουν ποιες είναι οι σεξουαλικές προτιμήσεις τους σύμφωνα με τα στερεότυπα που ισχύουν για τα άτομα αυτά ε, για τα LGDB δηλαδή για, τους, για τις λεσβίες, τους ομοφιλόφιλους κτλ. κτλ. Έχετε κάποια πρόθεση να κάνετε κάτι στο τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Σετόφσκι. Κύριε Σετόφσκι, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Κλοντ. Καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο να προφέρει κανείς ε, το όνομά μου. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Δεν το πρόφερα καλά. Είναι, είναι καλύτερα να με λέτε Τόμας. θα ήθελα να σας δώσω, θα σας, μπορώ να σας ζητήσω αυτά και γραπτός. Αλλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν ετέθη μέχρι στιγμής. Εγώ πήρα πληροφορίες ότι ένα τμήμα των μεταναστευτικών ρευμάτων αυτή τη στιγμή διακινείται υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού κράτους. Θα μπορούσατε να μας δώσετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το θέμα αυτό, ένα δεύτερο ερώτημα. έχουν στην Αίγυπτο 1.500 άτομα από τη Λιβύη με βίζες του συστήματος Σέγγεν. άτομα τα οποία όμως δεν είναι καθόλου καταγεγραμμένα στο σύστημα Σέγγεν. Δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία του Σέγγεν. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση όπου υπάρχουν κάτι τα οποία ξεκινούν αυτή τη διαδικασία, δίνουν προξενικές θεωρήσεις σε ασύλου και μετανάστες, οι οποίοι μετά έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τρίτο ερώτημα. Χθες, εγώ ήμουν έχω σταθεί συγητής για τα θέματα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχθη εκεί στη συζήτησή μας ότι η Frontex δεν συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη και δεν εφαρμόζει σωστά τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται βάσει του κανονισμού της Frontex. Μπορείτε να κάνετε κάτι για να βελτιωθεί λοιπόν αυτή η κατάσταση. Ε, thank you. Next is Tanya Fayon. Η Τάνια Φαγιόν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ρύθμιση των εφιών συνόρων και η σχετική νομοθεσία. Ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια και βεβαιότητα σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό. Εσείς είπατε ο ίδιος σήμερα ότι θα υπάρξει απόσυρση αυτή τη πρόταση και υπάρχει ανάγκη μιας μεταρρύθμιση. Εμείς έχουμε κάνει πολλέ συναντήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μαζί με άλλα θεσμικά όργανα έχουμε την ανάγκη να ελέγξουμε διάφορε τεχνολογίας και αυτό όμως θα απαιτήσει και μια, μια διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια. Το πραγματικό όμως ερώτημα είναι το εξής. Πώς θα λειτουργήσουν τα e, Εφή σύνορα υπό την έποψη του κόστους και της ε, προστασίας των δεδομένων. Θα χρησιμοποιηθεί λοιπόν στα σύνορα αυτά αυτό το σύστημα με τρόπο αναλογικό σε σχέση με τον στόχο που επιζητούμε να εφαρμόσουμε. Ποια θα είναι τα στοιχεία λοιπόν τα οποία θα, συνε... θα συλλέγονται στα σύνορα, ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά, ποιος θα είναι ο δικαστικός έλεγχος για αυτή την ε, συλλογή στοιχείων. Αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα, η πρόσβαση της δικαιοσύνης στα στοιχεία αυτά τα οποία συλλέγονται για τα άτομα στα σύνορα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορούμε να περιμένουμε μια νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο έτος, αν θα υπάρξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή των εφιών συνόρων. Ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη συνεχίζουν τη δράση τους. ώστε να έχουν οι δικαστικές αρχές πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και εδώ έχουμε πραγματικά αυτό το στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ κύριε Σκούλιαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις ε, που σχετίζονται με την έρευνα και διάσωση. Σχετικά με το πακέτο των έξυπνων συνόρων, χαιρετίζω την ε, πρότασή σας ε, να αποσύρετε την παλιά πρωτοβουλία και να παρουσιάσετε μια καινούρια. Να παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα πιλότο και πώς θα προχωρήσει το πακέτο αυτό. Στις 16 Οκτωβρίου στην συνεδρίαση μου είπα γιατί αυτό το έργο δεν μπορεί ε, να είναι διαχειρίσιμο με βάση τη νομική βάση της υπηρεσίας διότι παρακάμπτει τις αρμοδιότητες της δημοσιονομικές του Κοινοβουλίου και αποτελεί κακό προηγούμενο για το μέλλον. Η ερώτησή μου μπορείτε να διαβεβαιώσετε ε, ότι θα τηρηθεί πλήρως ο κανονισμός. Δεύτερη ερώτηση είναι για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση. Η υπηρεσία μετανάστευσης σκέφτεται ότι 3.000 πέθαναν προσπαθώντας να φτάσουν στα Ιταλικές ακτές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τα άτομα στην ανοιχτή θάλασσα να πεθαίνουν. Έχουμε τις εξωτερικά θαλάσσια σύνορα. Ήταν η εισήγησή μου. Ζητήσαμε ε, να συμμορφώνεται η Frontex με το διεθνές δίκαιο. Αλλά δεν έχουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση όπως και με το τεύτον, το πρόγραμμα τεύτον. Θα ήθελα να μου πείτε τι σκέφτεστε. Έχουμε λοιπόν δύο κανόνες. Έχουμε τις ευρωπαϊκές αποστολές που πρέπει να τηρούν τους κανόνες μας αλλά και τους εθνικούς. Είσαστε έτοιμος να θεωρήσετε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, ακόμα και τις επιχειρήσεις από τις εθνικές αρχές για έρευνα και διάσωση. Ε, θα αλλάξετε τον κώδικα αυτό των συνόρων Schengen. Σίλβι. Ναι, ήταν ενδιαφέρον αυτό το quiz αν θέλετε με τον βαμβαρδισμό ερωτήσεων. Μοιάζει με την ακρόαση που είχατε την προηγούμενη φορά. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για μια στρατηγική με συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούμε να συζητήσουμε και στο μέλλον. Δύο θέματα. Το ε, θέμα των εμπόρων ε, και τη εμπορίας ανθρωπίνων έντων γιατί δεν ακούμε περισσότερο να γίνεται λόγος για αυτά τα κυκλώματα και για τον κανονισμό Δουβλίνο 3, αν πρόκειται να υπάρξουν εξελίξεις για την κατανομή ε, των ετούντων, με βάση ποια κριτήρια θα μπορούσε να γίνει αυτή η κατανομή. Θα ήθελα, ε, πρωτού χάσουμε το θέμα, και ε, αυτό που είπε η Σίλβη Γκιόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε και πάλι να υποβάλουμε ε, σε αυτές τις ατελείωτες, ατέρμανες ερωτήσεις ε, τον Επίτροπο άλλη μια φορά. Δεν είναι νομίζω ο κατάλληλος τρόπος να προχωρήσουμε και στο μέλλον. Θα έχουμε θεματικές παρουσιάσεις με σημαντικά θέματα και τομείς. Αυτό είναι ουσιαστικό και για ε, νέα μέλη που δεν είναι συνηθισμένα σε, τέτοια, ε, σε τέτοιο τρόπο εργασίας ε, θα πρέπει να συνηθίσει ο καθένας, θα πρέπει να θέσει ο καθένας την ερώτηση που θέλει και μετά θα έχουμε πιο δομημένες συναντήσεις. Μετά τα όσα είπε η Σίλβη Γκιόν, επόμενη ερώτηση έρχεται από ζουλή Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Είναι το χάος στον κόσμο που δημιουργεί τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά και υπάρχει σαφής αντίφαση ανάμεσα στο γεγονός ότι μειώνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια ή την αναπτυξιακή βοήθεια με δραστικό τρόπο. Είναι, ε, υπάρχει ε, αν θέλετε, υπάρχουν εκπτώσεις, μειώνουμε κατά ένα τέταρτο την ανθρωπιστική βοήθεια. Σήμερα πληρώνουμε ίσως ε, για τους Σύριους πρόσφυγες. Τι θα γίνει αν δεν έχουμε πια χρήματα. Θα πρέπει να δράσουμε σε αυτό το επίπεδο, ίσως εσείς ως Επίτροπος και μετά για, με την φαντασία αν θέλετε. Η φαντασία είναι 3.070 που πνίγηκαν στην Μεσόγειο, άτομα που προσπαθούσαν να μπουν, να εισέλθουν στην Ευρώπη ε, και λιγότερο από 10 ε, τρομοκράτες. Είναι πολλοί, είναι 10 επιπλέον και θα πρέπει ε, να διορθώσουμε τα πράγματα. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτό το μείγμα μεταναστών, τρομοκρατών, μεταναστών, εγκληματιών. Είναι άνθρωποι που φεύγουν από το χάος και είναι ευθύνη μας. Έχω δύο ερωτήσεις πιο συγκεκριμένες. Ε, επίσης, ε, για θέμα φαντασίας, νομίζω ότι το γεγονός ε, της ανόρθωσης, της οικοδόμησης τείχων, όπως θέλουμε να κάνουμε στο Καλέ, νομίζετε ότι αυτό θα μειώσει τον αριθμό των θανάτων και τι σκέφτεστε για τον Κάμερον που θέλει να περιορίσει την ελευθερία κυκλοφορίας στο μέλλον. Και τέλος, θα ήθελα να μου πείτε για το τρίτον που τώρα και ένα μήνα λειτουργεί πόσα άτομα ε, βοηθήθηκαν ε, και πώς χρηματοδοτείται το πρόγραμμα αυτό και ποιος είναι ο συντονισμός του. Ναι, αυτό δείχνει πολύ καλά τα όσα είπα. Η απάντηση θα μπορούσε να απαιτήσει ε, μία ώρα απάντηση, Κάμερον κλπ. Ριάνο. Βλέπετε εδώ υπάρχουν ονόματα τα οποία δεν μπορώ καλά να προφέρω. Ελπίζω εν ευθέτω χρόνο να μπορώ να προφέρω καλά τα ονόματά σας. Όχι, νομίζω δεν θα μπορέσετε ποτέ. Είσαστε βέβαιος γι' αυτό. Μια ερώτηση. Θα ήθελα την αντίδραση του Επιτρόπου για τον λόγο την περασμένη Παρασκευή του David Cameron, του Βρετανού Πρωθυπουργού, για τη μετανάστευση και την μεταχείριση των μεταναστών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του Βρετανικού νόμου. Είχατε, μπορείτε να πάρετε το βραβείο για την πιο σύντομη ερώτηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Επίτροπε μας υπενθυμίσατε την αφοσίωσή σας στα θεμελιώδη δικαιώματα όπως και στην ακροασή σας. Χαίρομαι, αλλά θα σας κρίνουμε βάσει των πράξεων και όχι των λόγων, βάσει των συγκεκριμένων ε, δράσεων και μέτρων. Έχουμε όλο και περισσότερες εκθέσεις για τη μετανάστευση που καταγγέλουν την κατάσταση στην Μεσόγειο. Πάνω από 3.500 θάνατοι από την αρχή του χρόνου. Η οργάνωση μετανάστευσης γίνεται ότι είναι η πιο, η πιο επικίνδυνη ήπειρος ε, για τους μετανάστες είναι η Ευρώπη. Ποιοι είναι αυτοί που πέθαναν εδώ, αυτή είναι η ερώτησή μου. Είναι ουσιαστικά σήμερα πρώτον ε, Σύριοι, ε, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν, από την Αυγανία, από την Παλαιστίνη, όπως είπε η Ευαζολία, από το χάος του κόσμου. Άνθρωποι που δικαιούνται τη διεθνή προστασία. Μας λέτε ότι υπάρχει ένα κενό νομικό. Σας λέω όχι κύριε Επίτροπε, δεν υπάρχει κενό νομικό. Υπάρχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα είναι το Δουβλίνο 3. Μήπως δεν θα πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό χαίρεστε για το, ε, την διαδικασία του Χαρτούμ. Χαρτούμ ε, πρωτεύουσα μιας χώρας που είναι το Σουδάν, της οποίας χώρας ε, είναι, κατηγορείται ο, ο πρόεδρος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τι θα γίνει με μια διάσκεψη για τα μεταναστευτικά προβλήματα σε μια τέτοια χώρα. Οι πολίτες εκεί φεύγουν από μια εμπόλεμη ζώνη από ε, μια δικτατορία. Ε, νομίζω αντιμετωπίζουμε τα πράγματα από την ανάποδη. Τι θα κάνει η κυβέρνηση του Σουδάν, τη Ερυθρέας για να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, για να ενημερώσει για τους κινδύνους, για τους καταβλισμούς προσφύγων. Ξέρουμε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται και σας ζητά. Γιατί χαίρεστε για αυτή τη διαδικασία του χαρτούμ. Γιατί να πάμε να συζητούμε με αυτές τις χώρες που είναι δευτιαρμένες και που είναι υπεύθυνε ε, για την ε, εμπορία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κουτσίκα. Ε, the of in the Mediterranean and... Η κατάσταση για τους μετανάστες επιδεινώνεται όλο ένα και περισσότερο και ε, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους ετούντες άσυλο. Και προφανώς χρειάζεται μια ολιστική ε, αντιμετώπιση, να, υπά, να, βάλουμε μια προτεραιότητα στις διάφορες ε, ενέργειες που πρέπει να υιοθετηθούν και χαίρομαι που και για σας όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητα. Ήθελα να ρωτήσει πώς προτίθεται η Κομισιόν να κανονίσει θέματα επανεγκατάστασης. Υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση των προσφύγων ε, σε κάποιους καταβλισμούς. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δημοσιονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν ε, οι, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, πώς θα διαμορφωθεί αυτό το, το σύστημα επανεγκατάστασης αυτών των μεταναστών. Όχι, ο Επίτροπος με ρώτησε αν τελειώνουμε. Όχι, υπάρχουν ακόμα κι άλλοι. Όχι. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τον κατάλογο, συνάδελφοι. Μισοράγια Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά τον Επίτροπο και ε, πραγματικά ε, εύχομαι κάθε επιτυχία σε νέα θέση που έχετε αναλάβει. Κάποιες ερωτήσεις που ήθελα να θέσω έχουν τεθεί και θα ήθελα αν γίνεται να ε, υποβάλω κάποιες γραπτές ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Τώρα, τέλος πάντων, να πω όμως κάτι για, τους, ε, για την ελεύθερη ε, μετακίνηση και μετανάστες. Το, και το είπατε αυτό στην ίδια πρόταση. Για, όταν μιλάμε για ελεύθερη μετακίνηση, πρέπει να μιλάμε και για τους Ρωμά, που όμως δεν είναι άτομα τα οποία είναι μορφωμένα ή οτιδήποτε. Ε, αντιμετωπίζονται σαν ε, ζητιάνοι. Δεν είναι θέμα μετανάστευση το πρόβλημά τους. Θεωρώ ότι είναι προσβλητικό να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς ε, προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία αντιτίθεται στην ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων και που απελάβνουν κάποια άτομα. Κάτι άλλο. Σήμερα το πρωί μιλάγαμε για άτομα τα οποία ζητούν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τα δικαιώματά τους ε, έχουν ε, καταπατηθεί. Όταν, κυρίως όταν ζητάμε άσυλο. Ήθελα να ρωτήσω πόσο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα θέματα αυτά των ατόμων των οποίων τα δικαιώματα για αίτηση ασύλου δεν γίνονται σεβαστά. Άλλη ερώτηση. Θα πρέπει να έχουμε μια ανθρώπινη μεταναστευτική πολιτική. Αυτή η μεταναστευτική πολιτική που έχουμε τώρα είναι αντίθετη ε, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να βρούμε μια ε, σφαιρική λύση. Είχαμε το project Mare Nostrum πέρυσι. Ε, οι αιτούντες άσυλο δεν έρχονται εδώ για να διασκεδάσουν. Ε, προσπαθούν να ξεφύγουν από τον θάνατο. Ο κύριος Τζάκη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είσαστε αρμόδιος όχι μόνο για τα, για τα θέματα μετανάστευσης και εσωτερικών, αλλά είσαστε αρμόδιος και για τα θέματα ηθαγένειας. Γι' αυτό το ερώτημά μου αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Προβλητών. Εφέτος έχουμε προετοιμάσει μια αναθεώρηση του κανονισμού, κάναμε ακρόαση και προετοιμάσαμε μια έκθεση για το θέμα αυτό. Είναι γενικά γνωστό ότι η Κομισιόν δυσκολεύει αυτούς οι οποίοι καταθέτουν πρωτοβουλίες αυτού του είδους. Ως αποτέλεσμα, ο αντιπρόεδρος κ. Τίντερμανς είπε ότι υποστηρίζει το να δίδεται μια πολιτική απάντηση στις ε, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών. Ποια είναι η δική σας άποψη είναι το ερώτημά μου, πώς βλέπετε το μέλλον της ε, πρωτοβουλίας πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ιντεβέλτ, Σόφη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα και συγγνώμη που δεν ήμουν παρούσα στην αρχή όταν ε, ετέθηκαν ορισμένα θέματα για το ευρωπαϊκό PNR. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει εδώ πει ποτέ κατηγορηματικά όχι. Αλλά σε μια δημοκρατία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και οι, και οι διαδικασίες. Όταν προτείνεται μια νομοθεσία θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Σήμερα μετά από τόσα χρόνια συζητήσεων δεν έχουμε δει καθόλου στοιχεία για την αναγκαιότητα να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό PNR. Δεύτερον, το επιχείρημα της εναρμόνισης. Ξέραμε, προτού η Κομισιόν να προσπαθήσει να πει στα κράτη-μέλη να έχουν εθνικά συστήματα PNR ότι υπήρχε μοναχά ένα σύστημα, επομένως δεν έχει νόημα το επιχείρημα της ε, εναρμόνσης. Και σας υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών, οι βουλές των Κάτω Χωρών είπαν ένα καθαρό όχι στο σύστημα του, Ευρωπα... του εθνικού PNR. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδιο για να δημιουργηθεί το εθνικό σύστημα PNR στην Ολλανδία θα επιβάλλετε τώρα την υποχρέωση να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα και θα το περάσετε σε πείσμα του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Τέλος, λέτε ότι συνεχίζετε στην ίδια γραμμή όπως το παρελθόν. Εγώ νομίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει το ίδιο. Αν θέλετε λοιπόν να έχετε μια συμφωνία, θα σας πρότεινα να προωθήσετε με την ίδια στεναρότητα την οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα, όπως και για το Ευρωπαϊκό PNR. Εντάξει. Ακολουθεί. Η κυρία Σίσμαν. Ευχαριστώ. Σας χάνω. Είσαστε κάπου πίσω, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Κουσμάν. Κύριε Επίτροπε, η δική μου γενιά μεγάλωσε την εποχή που η το η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας λέγαν τότε για τα δικαιώματα, για την ευμάρεια, για όλα τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Αλλά κάποια στιγμή μεγαλώσαμε. Ήδη δεν πιστεύουμε αυτά τα οποία μας λένε. Το Ισπανικό κράτος έχει αυτή τη στιγμή φέρει στην πραγματικότητα τις περικοπές, την ανεργία. Οι νέοι έχουν πια πολλά προβλήματα να βρουν θέση εργασία, να έχουν ένα σπίτι, να έχουν μια οικογένεια, ένα μέλλον. Του μένει μονάχα η δυνατότητα να φύγουν από τι αιστείε του. Εκατοντάδε χιλιάδων έχουν φύγει και πολλοί άλλοι ετοιμάζουν τι βαλίτσε του. Και αυτό λόγω τη έλλειψη αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόσουν τα μέτρα ε, απέλασης από τις χώρες τους των ε, μεταναστών από τρίτες χώρες που τώρα θεωρούνται ότι είναι υπερβολικό βάρος. 4.812 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης εξεδίωξε το, Ευρω... το πρόσφατα και αυτό αφορά πια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ντέβιτ Κάμερον ενέκρινε αντίστοιχα μέτρα βάσει των οποίων μπορούν οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωση, οι οποίοι βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς θέση εργασία μετά από έξι μήνες να απελάβνονται. Στην Ευρώπη αρχίζουν να ορθώνονται τα εσωτερικά τείχη. Η οδηγία 2004-78 επιτρέπει τέτοιου είδους απελάσεις. Κύριε Πίτροπε, γνωρίζετε ότι αυτή η οδηγία παραβιάζει τη βασική αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας που είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τροποποιήσετε αυτή την οδηγία ή αντίθετα θα συνεχίσετε να επιτρέπετε τα κράτη-μέλη να απελάβουν Ευρωπαίους πολίτες και όχι μοναχά πολίτες τρίτων χωρών. Αυτό δεν οδηγεί παρά μόνο σε μεγαλύτερη ξενοφοβία υποσκάπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργεί όλο και μεγαλύτερα ρήγματα μεταξύ της Ανατολής, της Δύσης, του Βορρά και του Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Γιούνκερ είχε πει στην προεκλογική του εκστρατεία ότι όσον αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών, ε, η προάσπιση τους θα είναι μία από τις προτεραιότητες ε, του προγράμματός του. Αυτό αφορά το γεγονός ότι ε, η αίτηση για το άσυλο δεν θα γίνεται στην πρώτη χώρα, αλλά στη χώρα όπου ε, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να του χορηγηθεί το άσυλο και ε, θα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα οικογενειακής επανένωσης. Σαν αποτέλεσμα η Σουηδία πήρε διπλάσιο αριθμό αιτήσεων από την Ιταλία, η Γερμανία επίσης. Και όμως ε, στην Ιταλία είναι η χώρα που δέχεται τους περισσότερου ε, παράνο, ε, Εδώ τίθεται σε ε, κίνδυνο αν θέλετε ή μάλλον εμφανίζονται τα δύναμα στοιχεία και του συστήματος Σέγγεν και του συστήματος ε, της συνθήκης του Δουβλίνου. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, εσείς Ποια σχέδια έχετε, τι προτάσεις ε, θα υποβάλλετε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί που κάποιες χώρες είναι πολύ πιο ελκυστικές ε, ε, από κάποιες άλλες και που οι σε άσυλο πλέον έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την χώρα που θα υποβάλουν την αίτηση. Ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική για το άσυλο. Αλλά αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει κοινέ προδιαγραφές, κοινά πρότυπα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ε, ε, η οικονομική ε, κατανομή κατανομή του οικονομικού βάρους, τι θα γίνει ακριβώς. Η κυρία Κινίτσι, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μωράης, ευχαριστώ που δώσατε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα ακούσαμε για τη μετανάστευση. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα θέματα με αφορούν κυρίως όσον αφορά τους, ασυνόδευτα, τους μετανάστες ασυνόδευτα παιδιά και ε, τα σχετικά με τους ε, διακινητές. Ήθελα να κάνω πιο συγκεκριμένα μία ερώτηση για την ε, επιχείρηση τρίτων. Πριν από λίγες εβδομάδες στην, σε πέντε μέρες στο Αγκριτζέντο, στην περιοχή από την οποία προέρχομαι, έφτασαν 1.500 μετανάστες μέσα στα πλαίσια του project Mare εμφαρμόστηκε η επιχείρηση Τρίτονας. Ε, ήθελα να ξέρω πόσο καιρό περιμένετε να λειτουργήσει και ε, πώς βλέπετε να εκτιμάται η επιχείρηση αυτή, γιατί ούτως ή άλλως το μεταναστευτικό ρεύμα συνεχίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κατερίνα. Νομίζω ε, ούτω η αλλω το μεταναστευτικο ρευμα συνεχιζει συζήτηση, διότι ποτέ δεν υπήρξα σε μία συνεδρίαση όπου όλα τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν να θέσουν ερωτήσεις. Τώρα, ε, Μπορεί να δώσετε μια γενική απάντηση και αν λείπουν κάποια στοιχεία θα τα στείλετε και γραπτά, κύριε Επίτροπε. Αν υπάρξει και κανένα κενό, γιατί αυτό ήταν crossfire σήμερα πρέπει να πω, και για να κάνουμε και μια επισήμαση, ήταν πολύ πιο πιεστικό από ότι στο, στο hearing με την έννοια ότι ήταν και πιο ουσιαστικό. Εδώ γίνονταν δεν είμαστε για να ανοιχνεύσουμε τι προθέσει τη επιτροπή, αλλά να ακούσουμε τι θέσει τη επιτροπή Και έτσι δικαιολογώ πλήρω ε, και τα ερωτήματα και την πίεση που ασκείται. Πρώτα απ' όλα, θα επιτρέψετε να ξεκινήσω γιατί έχει σημασία επειδή εφήγει από αρκετού ότι οι αρχέ πάνω στι οποίε στηρίζεται η πολιτική του resettlement ε, είναι θεμελιώδης ε, για μας και εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για εκείνους που ζητούν, που επιδιώκουν νόμιμη είσοδο στην Ευρώπη. Είχα πει τότε, αν θυμόσαστε, ότι σε καμία περίπτωση η πολιτική μας δεν θα επιτρέψει να δημιουργηθούν όροι και συνθήκες απομονωτισμού της Ευρώπης. Είχα πει χαρακτηριστικά όχι σε μια Ευρώπη φρούριο. Και το επαναλαμβάνω και τώρα. Το ρησάδεμα λοιπόν είναι πολιτική priority, κυρία Κουντρίκα και γι' αυτό, όπως σας είπα, θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στην συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα στην Γενέβη. Ε, αναφέρθηκε η κυρία ε, Σοράλια στους ετούντες άσυλων. Ε, ελπίζω να, να σας έχω καλύψει με τα όσα έχω πει μέχρι τώρα. Σε ό,τι αφορά τον τρίτονα, το πρόγραμμα τρίτων, το οποίο πράγματι είναι σε εξέλιξη, Ήδη πρέπει να πω ότι μόνο θετικά αποτελέσματα δίνει. Είναι μία πιο ενισχυμένη ε, ε, μορφή της πολιτικής που ασκείται μέχρι τώρα. Ε, έχουμε 47 περιπτώσεις μέχρι στιγμής που έχουν καταγραφεί σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Όπως ξέρετε όμως η έρευνα και η διάσωση είναι μια εντελώς διαφορετική πολιτική και είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, ε, άφησα ένα κενό πριν στην απάντησή με την κυρία Χολμάγερ γιατί πρόλαβε ο χρόνος, αν και δεν είναι εδώ θα ήθελα να πω ότι ναι, είναι στις προτεραιότητές μας και αποτελεί αντικείμενο διαρκούς ε, συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση στη ρίζα του, του φαινομένου της ριζοστικοποίηση, του ριζοσπαστήμου του ραντικαλισμού. Σύντομα πρόκειται να ε, έχω και μία επαφή, σας το λέω με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης, ε, με ε, όλους τους εκπροσώπους των πολυμέσων που αυτόν τον καιρό παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, στην πληροφόρηση της διεθνούς κοινής γνώμης και όχι μόνο. Έτσι ώστε να βρούμε έναν τρόπο να περιορίσουμε την έκταση του φαινομένου και το κυριότερο να χτυπήσουμε στη ρίζα του ε, το ραντικαλισμό. Ε, κύριε Έγκελ, χαίρομαι που ε, αναφερθήκατε στην συνεργασία που ανατίσσεται ανάμεσα στους επιτρόπους. Ξέρετε, ε, στην αρχή το είδαμε αυτό σαν μια πρόταση πιλωτική, να δούμε αν θα δοκιμαστεί στην πράξη. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να γνωρίζει η Επιτροπή σας ότι η συνεργασία ανάμεσα στους επιτρόπους είναι εντυπωσιακά αλληλέγγυα. Δεν υπάρχουν ούτε τριβές, ούτε ανταγωνισμοί και εκεί όπου διασταυρώνονται οι αρμοδιότητες, γιατί ναι, είναι αλήθεια, είμαστε πάρα πολλοί αυτή τη φορά, βρίσκουμε ένα εσωτερικό modus operandi που μας επιτρέπει να καταλήγουμε σε συγκεκριμένες πολιτικές. Και πρέπει να σας πω ότι έχω τύχει ε, εντυπωσιακή ε, υποστήριξη από τους συναδέλφους μου που έχουν να κάνουν οι αρμοδιότητες με θέματα μετανάστευσης. Ε, πολύ ορθοδά αναφερθήκατε στην Ερυθρέα. Ξέρετε, στην Ερυθρέα υπάρχει ένα καθεστώς ε, διαβίου στρατιωτικές θητείες. Εκεί έχουν επινοήσει έναν πονηρό θα έλεγα τρόπο για να κρατούν υποκαθεστώς εχμαλωσίες τους ανθρώπους ε, ε, μέχρι το τέλος του βίου τους. Και βέβαια αυτό τους στερεί τη δυνατότητα να βρουν ε, δρόμους για να αναζητήσουν μια καλύτερη θέση στη ζωή. Θα σας πω όμως κάτι που συνέβη στα παρασκήνια των επαφών μας στην Ρώμη και πρωτήτερα γιατί χαιρέτησα τις πρωτοβουλίες Χαρτούμ ε, και Ραμπάτ. Πρώτα απ' όλα, το γιατί ονομάστηκε Χαρτούμ είναι μια άλλη υπόθεση. Εμεί το βρήκαμε αυτό. Το ότι ονομάστηκε Χαρτούμ δεν σημαίνει ότι αυτομάτως νομιμοποιείται και δικαιώνεται το καθεστώς σε αυτή τη χώρα. Αντίθετα, μάλιστα. Αλλά το Χαρτούμ υπάρχει σαν πόλη. Και επειδή εκεί έγιναν οι πρώτε συναντήσει, αυτό είναι. Δεν ονομάστηκε στη Ρώμη, δεν, δεν το βαφτίσαμε εμεί αυτό το πρόγραμμα Χαρτούμ. Η ουσία μα μας ενδιαφέρει. Στο περιθώριο αυτών των διεργασιών και διαβουλεύσεων, αν μου επιτρέπετε να. να... Γιατί να το αλλάξουμε όνομα τότε. Άμα εγώ δεν έχω κανένα αντίρρηση. Το η ουσία με ενδιαφέρει. Ε, θέλω λοιπόν να σα πω ότι στο περιθώριο είναι πάρα πολύ σημαντικέ συναντήσει με ε, εκπροσώπους όλων αυτών των χωρών και είμαστε συγκεκριμένοι εμείς τουλάχιστον ως προς τους όρους που θέσαμε σε αυτή τη ε, συζήτηση. Εμάς μας ενδιαφέρει η ανθρωπιστική πλευρά και βεβαίω το κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπτυξη υπό την έννοια ότι η Ευρώπη πράγματι διαθέτει πάρα πολλά χρήματα ώστε να βοηθούν αυτέ οι χώρες. Θέλω να σας πω ότι η πρώτη εντύπωση που αποκόμισε είναι ότι έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν μαζί μας. Και αυτό είναι θετικό. Θα υπάρξει δε και δεύτερη συνάντηση σύντομα. Η Ιταλική Προεδρία, πρέπει να το πούμε αυτό, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Ε, ο, ο κύριος ε, ε, Χουάν Φερνάντο Λόπεθ ε, Αγγιλάρ έθεσε μερικά ερωτήματα πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα για τα hot returns. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο εκτεταμένα αναφερθήκαμε σε αυτό. Ήταν η δεύτερη απάντηση που σας είχα δώσει. Δεν θα ήθελα να πω σε λεπτομέρειες ε, σήμερα. Ε, φυσικά ναι, ξεκάθαρη η απάντηση να δώσω, το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να παρακολουθούμε από κοντά όλες ανεξάρτητα τις χώρες στο βαθμό που αυτές πράγματι ανταποκρίνουν τις υποχρεώσεις τους. Ε, επίσης ε, για, την, ε, για την Βίζα, όπου είστε και εισηγητής όπως γνωρίζω, θα ήθελα να σας ζητήσω να το συζητήσουμε διεξοδικά και όπως είχαμε πει και στην κατηδία σύντομη συνάντηση που είχαμε στο Στρασβούργο, καλό θα είναι να κάνουμε μια συνάντηση. Βεβαίω θα είναι πολύ χρήσιμη, περισσότερο βέβαια για μένα, αλλά και για την χάραξη μια πιο συγκεκριμένη και πολιτική. Ο... Δεν θυμάμαι και εγώ το, το επώνυμο, μας είπα να τον λέμε Τόμας, αλλά ο Τόμας ε- έθεσε κάτι πριν ε, σχετικά με τη Frontex. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή υπήρξε ένα κενό στην ε, διερμηνία και δεν ε, ε, συνέλαβα, δεν έλαβα το πρώτο σκέλος ερώτηση. Ως προς την Frontex όμως, πρέπει να σας πω ότι αυτό το πρόγραμμα έχει αποδειχθεί επιτυχές. Θέλει βελτίωση, θέλει ενίσχυση, θέλει αναμπάθμιση. Ποια είναι λοιπόν η πολιτική μας θέση. Θα την ενισχύσουμε την, ε, την Frontex. Γιατί πράγματι ε, δημιουργεί μια ομπρέλα προστασίας την ίδια στιγμή όμως πέραν από του βασικού σκοπού που είναι η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων που επιτρέψτε να σας πω ότι κάποτε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και αυτή την έννοια των ευρωπαϊκών συνόρων αλλά δεν είναι για την σημερινή μας συζήτηση ε, προσφέρουν στην πράξη χρήσιμες ε, υπηρεσίες και ανθρωπιστική βοήθεια. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί δείχνουν ότι δεν εξαντλείται η Frontex μονάχα στη συγκεκριμένη αποστολή της αλλά πηγαίνει ακόμα παραπέρα. Η κυρία Τάνια Φαγιών αναφέρθηκε στα smart borders. Βέβαια έλειπε στην αρχή που ε, αναφέρθηκα εκτενώς. Ε, είπα όμως ότι το αποσύρουμε ε, και χαιρετίστηκε αυτή μας η θέση. Θα επανέλθουμε όμως με μια καινούργια ολοκληρωμένη πρόταση. Κατά τη διάρκεια της περίοδου να ξέρετε, να ότι θα λάβω πολύ σοβαρά υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που έχουν, που έχουν γίνει. Ε, μισό λεπτό. Ε, δεν ξέρω αν με ρώτησε κάτι παραπάνω κυρία ε, ε Σε ό,τι αφορά ε, ε, τον κύριο Κοέλιο. Κύριε Κοέλιο, έχετε δίκιο. Δεν είναι όμως pilot project, δεν είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Όπως ακούσατε, είναι η τελική φάση η δεύτερη της διαδικασίας θα ακολουθήσει μετά την μελέτη που περιμένουμε και η οποία είναι σε ε, εξέλιξη. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται υπό την επίβλεψη της Επιτροπής. η κυρία Σιλβί Γιώμα αναφέρθηκε στην καταπολέμηση των σμάγκλες και έκανε και μία παρατήρηση ε, ε, πλέον για την συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτήν την ε, εγκληματική δραστηριότητα αν δεν αναπτύξουμε συνέργειες ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Και όπως είπα πρωτήτερα και επαναλαμβάνω και τώρα, η ανταπόκριση ακόμα και των transit countries είναι θετική. Και σε αυτή ανάλυση και αυτές θίγονται από την δραστηριότητά τους. Ε, το είπα και πριν και επανέρχομαι στην κυρία Εύα Τζολή. Δεν πιστεύω στην Ευρώπη Φρούριο και σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον είναι μια δέσμευση που έχω αναλάβει απέναντι σε εσά και απέναντι κυρίως στην συνείδησή μου. Τώρα, έγινε αναφορά στις δηλώσεις του κυρίου Κάμερον. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Απλώς θα ήθελα να σα πω ότι πότε λαμβάνουμε ο κύριος Κάμερον αναφέρθηκε στην ε, ελεύθερη κίνηση των Ευρωπαίων πολιτών όχι μεταναστών από τρίτες χώρες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, και αυτό είναι μια κατάκτηση της Ευρώπης, ελέγχθη πρωτήτερα και θα συμφωνήσω απόλυτα με όποιους το έδωσα, δεν μπορούν να θεωρούνται μετανάστες μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είμαι βέβαιος ότι το θέμα των δηλώσεων του κ. Κάμερον θα συζητήσετε στην επικοινωνία που θα έχετε με την κυρία ε, Ζούρβα, τι οποίε και η αρμοδιότητα γενικότερα είναι αυτά τα ζητήματα. Τώρα, για το Δουβλίνο. Το είχαμε πει και παλιότερα. Το Δουβλίνο καθημερινά δοκιμάζεται στην πράξη. ω προ κάποια σημεία του λειτουργεί. Είναι under monitoring. Το παρακολουθούμε. Έγινε μια προσπάθεια, γνωρίζετε, με την αναθεώρηση του άρθρου 33 για τη βελτίωση τη λειτουργία του. Παρόλα αυτά, εγώ θα σα πω, ότι από την ώρα που ε, στην πράξη δοκιμαζόμενο το Δουβλίνο κριθεί ότι δεν ανταποκρίνεται με επιτυχία στους σκοπούς που εκλήθη να υπηρετήσει, ναι, θα προχωρήσουμε σε αλλαγές. Αλλά όλα αυτά, εφόσον προκύψει ανάγκη, γιατί τώρα δεν έχει τέτοιο ζήτημα, θα γίνει σε συνεργασία ε, μαζί σας. Η εμπειρία και οι παρατηρήσεις σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε μένα. Τώρα για τους Ρωμά. Θυμίζω Μιας και αναφερθήκατε στους Ρωμά, οι Ρωμά δεν, δεν, είναι, δεν είναι migrants, είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Και νομίζω ότι από μόνο του αυτό απαντά στο σημείο που δείξατε. Για την ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, γνωρίζετε ότι αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρτοφυλακίου του κυρίου Τίμερμανς. Διασταυρώνεται όμως και με το citizenship. Ε, σύντομα ε, θα ζητήσω από τον Πρόεδρο να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα της ηθαγένειας. Ξέρετε, προσεθέθησε το χαρτοφυλάκιό μου στην τελευταία στιγμή και πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν είχα καν τον χρόνο για να μελετήσω σε βάθος όλες, ε, όλες τις φάσεις και τις πτυχές αυτού του τόσο σημαντικού ζητήματος που έχει να κάνει και με την ευρωπαϊκή ταυτότητα και με θεσμικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πάντως είναι πολύ σημαντικό θέμα και εγώ θα επανέλθω ε, ε, για να σας ενημερώσω. Ε, δεν νομίζω ότι έχω ε, τίποτα άλλο να προσθέσω. Α, ε, ναι, το, για το PNR ε, έγινε πάλι μια αναφορά. Δεν είσαστε στην αρχή, λυπάμαι που δεν είσαστε εδώ, αλλά θα το συζητήσουμε σίγουρα πάρα πολλές φορές. Εγώ προσωπικά εκτιμώ και έχω πιστεί ότι υπάρχει ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό PNR. Το απήντησα προλίγο νομίζω και στην κυρία Σπινέλη, αν δεν κάνω Είναι μια ξεκάθαρη θέση. Το πώς αυτό όμως θα λειτουργήσει και πώς αυτό θα προστατεύει στην πράξη τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κάτι το οποίο έχουμε λάβει σοβαρότατα υπόψη, πάντοτε όμως έχοντας κατά νου ότι πρέπει να δημιουργήσουμε και τις όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή η λειτουργία της ε, κοινωνίας και κυρίως σημαντικών τυχών της που έχουν να κάνουν ε, κυρίως με τις αερομεταφορές. Γνωρίζετε και τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί τον τελευταίο καιρό και από τους άμεσα ε, ενδιαφερόμενους. Ε, επίσης για τον κύριο Κινίτσι θα ήθελα να πω ότι ο τρίτον πώς, κυρία. κυρία Κινίτσι ο τρίτον, ο τρίτον δεν αντικαθιστά το πρόγραμμα Mare Nostrum ε, στηρίζει την ε, δράση των κρατών μελών για προστασία, για προστασία ε, συνόρων. Ε, τελειώντας θα ήθελα να σας πω ότι όλο και περισσότερο αναπτύσσουμε ε, πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην καλλιέργεια της απαραίτητης αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Διότι μεταναστευτική πολιτική Χωρίς ε, την ε, απαραίτητη αλληλεγγύη δεν θα μπορέσει ποτέ να επιτύχει και η αλληλεγγύη πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη. Πονηρές πολιτικές που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν και που αποβλέπουν στο να μεταθέτουν εντός εισαγωγικών το βάρος από τη μία χώρα στην άλλη δεν είναι σωστό ούτε είναι δίκαιο. Πρέπει να διασταυρώσουμε την αλληλεγγύη με την ευθύνη όμως των κρατών μελών και πρέπει να σας πω ότι μία από τις πρωτοβουλίες που σήμερα θα αναπτυχθούν είναι και σε επίπεδο συμβουλίου να γίνει μία συζήτηση έτσι ώστε ο καθένας να επιμεριστεί και να αναλάβει το μέρος ευθύνης του αναλογή. Πάντοτε κάτω από τις βασικές αρχές που διέπουν την ευρωπαϊκή ε, πολιτική και που έχουν να κάνουν και με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κοινοτικού κεκτημένου και του χρέους μας να δημιουργήσουμε περιβάλλον ε, ανθρώπινο για όλους τους πολίτες της Ευρώπης αλλά και για όσους επιλέγουν να περάσουν τις πόρτες της Ευρώπης και να ενταχθούν στις κοινωνίες μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Όσο είσαστε ακόμα εδώ μου είπανε τα μέλη ότι ο, ότι ο Μπαρό ο οποίος υπήρξε Ζακπαρό που υπήρξε μέλος της Επιτροπής στην προηγούμενη Επιτροπή πέθανε και πολλά μέλη έχουν τονίσει ότι πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στον μετελθόντα Επίτροπο ο Ζακπαρό Και μετά από 46 ερωτήματα δεν ξέρω αν έχει καταστεί δυνατό ο κύριο Επίτροπο να απαντήσει σε όλους ικανοποιητικά. Αλλά είναι η μόνη ευκαιρία που έχουμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τους έξι επιτρόπους με τους οποίους εμπλέκεται η Επιτροπή μας δεν πρόκειται να κάνουμε μια τέτοια διοργάνωση και πάλι. Στο μέλλον θα έχουμε μια πιο στοχευμένη εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα όπως είναι το PNR, τα e, σύνορα, η νόμιμη μετανάστευση η Μεσόγειος κτλ. Έτσι θα λειτουργήσουμε το μέλλον. Θα εστιάσουμε λοιπόν περισσότερο σε συγκεκριμένα θέματα, ώστε να έχουμε πιο λεπτομερείς ε, απαντήσεις και πιο στοχευμένο διάλογο. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό τα νέα μέλη και τα παλιά μέλη που γνωρίζουν καλύτερα τα θέματα αυτά να έχουν την ευκαιρία να γίνει αυτή η ευρεία συζήτηση για να αντιμετωπίσουν όλα τα ζητήματα που είναι στην ε, αρμοδιότητα του κ. Αβραμόπουλου. Νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα είναι οι επόμενες επαφές μας τόσο σκληρές όσο οι ακροάσεις των Επιτρόπων και χαίρομαι που οι βουλευτές της Επιτροπής μας μπόρεσαν να θέσουν και να λάβουν απαντήσεις σε, στα ερωτήματά τους. Η επόμενη συνάντησή μας θα εστιάζει σε κάποια συγκεκριμένα θέματα αν θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ θα ήθελα να πω, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, θα προτιμούσα να είχα πιο θεματικού χαρακτήρα συναντήσεις, θα ήταν ουσιαστικότερες και θα με βοηθούσαν και εμένα. Ευχαριστώ λοιπόν τα μέλη για την ε, υπομονή τους. Ευχαριστώ τους συντονιστές και τα μέλη που έθεσαν ερωτήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για το γεγονός ότι δείξατε υπομονή και ακόμα και για αυτούς που δεν πήραν την απάντηση που θέλανε ενδεχομένω. Σας ευχαριστώ για την πειθαρχία που δείξατε. Μπορέσαμε να δώσουμε σε όλους το λόγο και να πάρετε απαντήσεις. Ακόμα και δεν ήταν η απάντηση που θέλετε. Σας ευχαριστώ πάλι κύριε Επίτροπε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία σας και προσβλέπουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ. Um, Συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, που αφορά την αντιμετώπιση των παιδιών και τις δικονομικές εγγύσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι κατηγορούμενοι στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, δημοσιοποιήσει ένα, μια, οδηγία για το, μια πρόταση για οδηγία για την ε, ε, ενίσχυση των εγγύσεων για τα παιδιά που είναι υποπτή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών. Ήδη από το Μάρτιο του 2014 δημοσιεύθηκε ένα έγγραφο εργασίας από τον προηγούμενο εισηγητρή που είχε υιοθετήσει μια γενικότερη προσέγγιση. Η Κατερίνα Κινίτσι είναι τώρα αυτή η οποία αναλαμβάνει ω εισηγήτρια. Είχαμε και μία πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση για το θέμα αυτό και ε, επίσης και για τα θέματα της ε, ε, χορήγησης νομικής βοήθειας. Κυρία Κινίτσι, έχετε το λόγο. Το τεκμήριο Για το τεκμήριο παινίας, πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, κυρία Κινίτσι, έχετε το λόγο. Κατερίνα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη που ανέλαβα αυτό το θέμα, αυτό το φάκελο, ε, σαν την το πρώτο καθήκον που αναλαμβάνω ε, ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα τα, το οποίο με απασχόλησε εκεί στην, Ιταλία και στο τμήμα ανηλίκων και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, για τους ανήλικους πάντα. Ε, η εμπειρία μου αυτή μου χρησιμεύσε στην ε, αξιολόγηση και στην εκτίμηση της οδηγίας, διότι είχαμε τον τρόπο αυτό ένα είδος μπούσολα, το οποίο έπρεπε να, μπούσουλα, το οποίο έπρεπε να ακολουθήσω για να καταλάβω, να αξιολογήσω καλύτερα την οδηγία. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο ουσιαστικές απαιτήσεις ε, στις οποίες προσπαθεί να δώσει μία ε, απάντηση η οδηγία. Το ένα είναι ότι να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των ανηλίκων, το δεύτερο είναι να ε, σεβαστούμε και την όλη δικονομική διαδικασία στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στις χώρες μέλη. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία Ε, εξαρτάται και από την ε, ευθύνη του υποκείμενου ε, και του, του υπεύθυνου για, την, για το αδίκημα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα άτομο, το οποίο, για ένα υποκείμενο το οποίο είναι ευάλωτο, το οποίο είναι ευάσθητο, ευαίσθητο. Γι' αυτό και η οδηγία την οποία συζητάμε σήμερα θέτει κάποιες σημαντικές εγγύησεις για την προστασία του υποκειμένου αυτού. Όπως θα θυμόσαστε ότι η οδηγία για, για τους ανήλικους εντάσσεται παράλληλα με τις άλλες ε, προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην, ε, ε, στο όλο πλαίσιο για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων ή αυτών οποίων ερευνώνται για την στα πλαίσια των ποινικών διαδικασιών. Ήθελα να πω ότι σύμφωνα με τις άλλες οδηγίες του πακέτου, η οδηγία για τους ανήλικους είναι πιο συγκεκριμένη, διότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περιορίζεται απλώς και μόνο στις ε, δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών. Από την άλλη πλευρά, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι ευρύ, διότι σε αντίθεση με άλλα θέματα που αφορούν μόνο μία πτυχή των δικονομικών εγγύσεων, η οδηγία για τους ανήλικους αναφέρει ε, έναν ολόκληρο κατάλογο δικαιωμάτων που αφορούν τους ε, ανήλικους που είναι ύποπτοι κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και έχουμε να κάνουμε με ένα, ε, σύνολο άχιστων ε, προδιαγραφών που είναι απαραίτητες να γίνουν σεβαστές για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των ε, ανηλίκων. Επομένως, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο σωστής δικονομικής διαδικασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των παιδιών, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή λείπει. Γι' αυτό ακριβώς ο λόγο θα ήθελα να πω ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές αυτή τη στιγμή. Ε, ε, υπάρχουν εκατομμύρια ανήλικοι οι οποίοι εντάσσονται ε, στο, στις ποινικέ διαδικασίες στην, στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να εναρμονίσουμε την, τις νομοθεσίες έτσι ώστε οι διαφορές αυτές που υπάρχουν να εξομαλυνθούν. Ήθελα να πω ότι εξέτασα ε, τον, την πρόταση του προηγούμενου εισηγητή, την οποία έχει εξετάσει και η Κομισιόν και συμμερίζομαι ε, την γενική προσέγγιση της οδηγίας και το βασικό περιεχόμενο. Ε, πιστεύω ότι η οδηγία αυτή έχει συνταχθεί με την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό βήμα ε, όσον αφορά την ε, αναγνώριση των δικαιωμάτων των ανηλίκων που έχουν εμπλακεί σε αυτές τις ποινικέ διαδικασίες. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, μία από τις βασικές πτυχές πτυχές της πρότασης της Κομισιόν είναι ε, η, νομική αρρωγή. Ε, είναι ένα δικαίωμα που έχει το παιδί, ε, αυτό το ευεργέτημα παινίας, το οποίο δεν μπορεί να αποποιηθεί. Είναι μια εγγύηση η οποία δεν αφορά μόνο την ποινική διαδικασία, αλλά έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει την εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων που έχει το παιδί. Ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ε, τις εγγύησει ε, ε, όσον αφορά την ανάκριση, την, το ότι ο, ο ανήλικος συνειδητοποιεί πλήρως την διαδικασία της οποίας αποτελεί ένα κομμάτι πρέπει να συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο ρόλος όλων όσων έρχονται σε επαφή μαζί του και οι προβλέψεις σχετικά με την στέρηση της ελευθερίας του ε, ανήλικου όταν η, η ποινή της φυλάκισης θα πρέπει να ε, αποτελέσει την ίστατη ε, ποινή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται εναλλακτικές ποινές. Αυτά είναι τα, αυτό είναι το βασικό, το βασικό περιεχόμενο της οδηγίας το οποίο, το οποίο συμμερίζομαι. Προσπαθώ να είμαι σύντομη, αλλά τέλος πάντων ε, πρέπει να σας πω ότι μέσα στα πλαίσια των τροπολογιών προσπάθησα να ενδυναμώσω, να ενισχύσω τις εγγύσεις που ήδη υπάρχουν. Στα πλαίσια των διευρύνσεων που έγιναν σε σχέση με την αρχική πρόταση, να υπενθυμίσω κυρίως ε, την πιο γενική ε, διάταξη που αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, το άρθρο 2, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής ε, τα άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους, δεν είναι 21 όμως ακόμα και το, το το έχουν διαπράξει πριν ε, συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικία τους. Θα πρέπει να εγγυηθούμε ε, τα, τα δικαιώματά του τη στιγμή που διέπραξε το αδίκημα, δηλαδή τη στιγμή που δεν ήταν ε, σε πλήρη γνώση του τι έκανε. Τώρα για κάποια άλλα δικαιώματα, το 41, 42, 43 που αφορούν το δεύτερο, δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 που αφορούν τα, την κράτηση των ε, ανηλίκων. Πρέπει σε περίπτωση φυλάκισης ε, οι δομές να είναι κατάλληλες, η μεταχείριση να είναι κατάλληλη και ε, τα άτομα τα οποία, και τα ανήλικα τα οποία κρατούνται πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση και με τα συμπεράσματα, γιατί όπως σας είπα θέλω να είμαι σύντομη, μέσα στα πλαίσια του άρθρου 3 θεωρήσαμε ότι, το να, ότι έπρεπε να εισάγουμε ε, την διάταξη που λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν παραμένουν αμφιβολίες, ε, αυτές οι αμφιβολίες θα πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση για την γωνιακή ευθύνη ε, πρέπει να ε, πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη κάποιος από τους δύο γονείς και θα πρέπει να δούμε στην περίπτωση που δεν υπάρχει ε, γωνιακή ευθύνη, ποιος θα είναι ο ενήλικας, ο οποίος θα αναλάβει την ε, ευθύνη για τον ανήλικο. Δύο διευκρινήσεις περαιτέρω. Την εισαγωγή μιας νέας παραγράφου στην αρχή του άρθρου 12 που αναφέρεται στην, ε, στην περίπτωση στέρησης της ελευθερίας και την εισαγωγή ενός νέου άρθρου στα, για τα μέσα προσφυγής πέραν αυτών που προβλέπονται στην οδηγία. Και αυτό σε αναλογία με τα όσα προβλέπουν οι άλλες οδηγίες του πακέτου. Σταματάω εδώ, κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο επειδή δεν μου δώσατε, ε, μου δώσατε συγκεκριμένο χρόνο, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με άκουσαν με προσοχή γιατί και ε, από πλευρά τους ε, αναγνώρισα αυτή την ευαισθησία ε, για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους θέματα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Κατρίν. Όταν έχουμε ένα συνάδελφο που γνωρίζει τα θέματα και εκπονεί την έκθεση στην αντίστοιχη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ήμουν στην ακρόαση του Νοεμβρίου και δεν θα ήθελα να είμαι στην θέση αυτή που προσπαθώ να επιταχύνω τη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, όπως ήταν και η ακρόαση της 11ης Νοεμβρίου. Αλλά πήραμε τόσο πολύ χρόνο με την ε, συνάντηση με τον κύριο Επίτροπο και αυτό ήταν ε, κάτι που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε και ακολουθεί ένα θέμα το οποίο πρέπει να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Θα ήθελα τώρα να ξέρω Ποιοι σκιώδεις εισηγητές θέλουν να λάβουν το λόγο. Ξέρω ότι ο κ. Τζάκη θέλει να λάβει το λόγο. Μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχει κάποιος άλλος σκιώδης ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Θα μου το πείτε τώρα. Η Σίλβη Ιβών, ναι, θέλει να λάβει το λόγο. Κλείνω λοιπόν τον κατάλογο, παρακαλώ, δεν ξέρω αυτό είναι πρόβλημα. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τζάκη, ο οποίος είναι ο σκιώδης του ΕΛΚ. Παρακαλώ να είστε όσο μπορείτε πιο σύντομοι. Γιατί πράγματι έχουμε πίεση χρόνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ουγγρικά. Θέλω να χαιρετήσω το σχέδιο έκθεση. Είναι πολύ καλή εργασία. Πιστεύω ότι στην Επιτροπή μας υπάρχει μια συμφωνία διαπαραταξιακού χαρακτήρα. Θέλουμε να προχωρήσει αυτό το έγγραφο και να έχει υψηλή ποιότητα. Είναι αναπόφευκτο ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τα τραύματα τα οποία υφίστανται τα νεαρά άτομα αυτοί οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την ηλικία του το 18 και εκεί είναι δύσκολο πολλές φορές να έχουμε από τα έγγραφα του πεδίου την πραγματική του ηλικία, θα πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Πρέπει να βρούμε και μια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι ο καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Αν έχουμε ενώπιον μας ένα ανήλικο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η ανήλικη είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, κάθε περίπτωση είναι χωριστή. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια κατά περίπτωση αξιολόγηση της κατάστασης. Θα πρέπει να δώσουμε ε, έμφαση στην ε, οριμότητα του ατόμου αυτού, στην κατάσταση της υγείας του, στην κατάσταση την οικογενειακή και κοινωνικο-οικονομική. Βρισκόμαστε τώρα στην αρχή μιας διαδικασίας, στα επόμενα Δήματα θα έχουμε τις προτάσεις τροπολογιών που θα κατατεθούν. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μαζί με την κυρία εισηγήτρια και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία εν ώψη των, διαπραγματεύσεων που πρέπει να διεξαγάγουμε με το Συμβούλιο. Το οποίο σημαντικό είναι να μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να προστατεύσουμε τα παιδιά τα οποία βρίσκονται υπό ανάκριση ή κάτω από υποψία να τους προστατεύσουμε. Και θέλω λοιπόν αυτό να τονίσω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τζάκη. σας ευχαριστώ για την συντομία σας Η Λάουρα Φεράρη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Κινίτσι. Την συγχαίρω κιόλα για την ε, και τον τρόπο που και το και τις γνώσεις που έχει για να συντάξει την έκθεση αυτή. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για τις αλλαγές που έχουν γίνει, τροπολογία 14 για το άρθρο 21 που διευρύνεται η δυνατότητα παρουσίας του δικηγόρου αλλά και κάποιου κηδεμόνα έτσι ώστε να μην παραμένει απροστάτευτος ο ανήλικος ή για την διεύρυνση των δικηγόρων οικονομικών εγγύσεων στα άτομα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικία τους και για επίσης για τη διευκρίνηση των όρων σύλληψης. Λοιπόν, ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Η κυρία Σιλβί Κάουφμαν. Ευχαριστώ και εγώ ήθελα να λάβω το λόγο γιατί θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, έκθεσή της. Την είδα είναι πολύ καλά διατυπωμένη θέλουν να ενισχύσουν τα δικαιώματα των παιδιών και κάτι άλλο που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι στο άρθρο 3 αναφέρει η συγκήτρια ότι όταν δεν ξέρουμε πώς, σε τι, ποια ηλικία βρίσκεται πραγματικά ένα παιδί, τότε η αμφιβολία πρέπει να είναι υπέρ του ανήλικου. Γι' αυτό ελπίζω ότι θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η έκθεση και να αποσπάσει μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού μια πολύ σωστή αντιμετώπιση και απάντηση από μια πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήθελα κάποτε να το πω αυτό, Σιλβί Ιβόν. Μου έδωσε την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες τώρα έχει αλλάξει 6 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Το υπενθυμίζω στους συναδέλφους για όσους θέλουν να καταθέσουν σχετικές τροπολογίες. Μήπως μπορείτε να με συμβουλέψει τώρα η γραμματεία. Πόσο χρόνο έχουμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Κομισιόν και στην Προεδρία. η πίεση χρόνο έχουμε. Μεγάλη λέει. Νεύων η γραμματεία. Πολύ μεγάλη ή μεγάλη. Καλά. Δεν είναι τραγικά τα πράγματα. Η Κομισιόν πρώτα. Αν μπορεί σε ένα λεπτό να σε δύο λεπτά ίσως να λάβει το λόγο. Αν μπορείτε να εστιάσετε σε αυτά που είπε η συγγήτρια φυσικά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος Κομισιό θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια για την, ε, το σχέδιο έκθεσης που θα επιτρέψει περαιτέρω πρόοδο σε αυτά τα σημαντικά θέματα. Πράγματι χαιρετίζουμε και καλωσορίζουμε ιδιαίτερα αυτή την έκθεση η οποία διατηρεί μια φιλόδοξη και πλήρη προσέγγιση όπως και η πρόταση της Κομισιόν και λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα δικαιώματα. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες όπως ε, τόνισε η κυρία Κινίτσι το πιο σημαντικό ερώτημα, η πιο σημαντική πρόνοια είναι η υποχρεωτική αρρωγή. Το τεκμήριο για τους ανήλικους και μας επιτρέπει να κρατήσουμε την αρχική μας φιλοδοξία. Η κατά περίπτωση προσέγγιση σε εξαιρέσεις προς το συμφέρον του παιδιού είναι σημαντικές για να μπορέσουν να μην χρησιμοποιηθούν κριτήρια αναλογικότητα, τα οποία κινδυνεύουν να είναι ιδιαίτερα σαφή. Θέλω εκτέλους από την πλευρά της Κομισιόν την ε, θέλησή μας να βοηθήσουμε την εισηγήτριά σας και την Επιτροπή σας ώστε να προχωρήσει ο, η εκπόνηση εκθέσεως και ο τριγωνικός διάλογος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, την κυρία Κινίτσι, για αυτή την έκθεση, την αρχική έκθεση, την οποία υποδεχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι από πλευρά του Συμβουλίου μπορώ να πω ότι οι στόχοι που έθεσε η συγγήτρια και που αποτέλεσαν την κατευθυντήρια γραμμή της έκθεσης είναι οι ίδιοι στόχοι που ακολούθησε και το Συμβούλιο. Να υπάρξει μια ισορροπία δηλαδή ανάμεσα στην ενδυνάμωση, στην ενίσχυση των δικονομικών εγγύσεων για, τα, για τους ανήλικους, γιατί είναι ευαίσθητα και ευάλωτα άτομα και τον στόχο των δικονομικών διαδικασιών, διότι... η οι ποινικέ διαδικασίες έχουν σαν στόχο να εντοπίσουν ποιο είναι υπεύθυνο για ένα συγκεκριμένο αδίκημα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα δικαιώματα των θυμάτων που θέλουν να ξέρουν ποιο είναι υπεύθυνο. Ναι και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας να πω για το, τις αμφιβολίες όπου ανακούστηκαν δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω ήδη τον Ιούνιο το Συμβούλιο ασχολήθηκε με την νομική αρρωγή και ήθελα να υπενθυμίσω ότι για τα θέματα του individual assessment υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου, μία θέση του Συμβουλίου που προσεγγίζει αυτή του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί ένας, ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής Υπάρχει μια κάποια απόσταση ακόμα, αλλά επειδή είναι κοινέ οι προσδοκίε μα όσον αφορά το κείμενο, ε, ε, όπω είπε και η συγγήτρια η κυρία Κινίτσι, ε, νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε το έργο μα. Επίση, όσον αφορά του χρόνου, θέλουμε να ξεκινήσουμε τον πιο γρήγορα τη συνεργασία μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το τέλος της θητείας ε, ήταν, λειτουργήσε εναντίον μας, αλλά τέλος πάντων είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, για να διευκρινιστεί και η διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει όλες οι αντιπροσωπείες να συνεργαστούν έτσι ώστε να καταλήξουν σε ένα πιο γρήγορα σε ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να γίνει δεκτό από όλα τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, σας είπα ποια είναι η νέα προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ. Ευχαριστώ Κατερίνα, ευχαριστώ τους συναδέλφους. And... Λοιπόν, είναι 6 παρατέταρτο. Και περνάμε στα θέματα, στο θέμα και κλεισμένων των θυρών. Άρα όλοι όσοι δεν έχουν την... Ε, δεν μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα, καλό είναι να αποχωρήσουν. Όσο τον πιο γρήγορα και πιο ήσυχα μπορείτε.